La Ξεκινάει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα παρακαλέσω όσους είναι όρθιοι και συζητάνε να έρθουν να καθίσουν επειδή ήδη έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση και η συνάντησή μας έχει πολλά θέματα και είναι και πολύ σημαντική. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε χρόνο να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να καλωσορίσω τα 25 μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που εκπροσωπούν σήμερα 13 χώρες της Ένωσης. Αποφελούμε λοιπόν της ευκαιρίας για να στήσω συγγνώμη για τη χώρα μου για την οποία θα έπρεπε να είχαμε τρία μέλη, τρεις εκπροσώπους, αλλά σήμερα είχα μια πολύ σημαντική ψηφορία στο Κοινοβούλιο και δεν μπόρεσαν να έρθουν. Βεβαίω θα του μεταφέρω έτσι μια σύνοψη των εργασιών μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η έκθεση για την ενιαία αγορά όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που εγκρίθηκε την 7η του Σεπτέμβρη ζητούσε μια καλύτερη επικοινωνία σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα την κυρία Μαρλή Σπίσιντζέρα, εκπρόσωπο τη Αλβετία, συγγνώμη αν έκανα λάθο το όνομά σα, και τον εκπρόσωπο τη Νορβηγία, τον Τέρλ Σβίρκομ. Βεβαίω, θα ήθελα να καλωσορίσω και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Ενιαίας Αγοράς εσωτερική συγγνώμη αγορά. Βλέπω και κάποιοι να λείπουν. Φαίνεται ότι παρακάθισαν στο μεσημεριανό γεύμα και θα χάσουν σημαντικέ έτσι σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι υπό το φω τη ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και μετά βεβαίω από την παρουσία των εκπροσώπων των ε, κοινοβουλίων των χωρών μελών θεωρώ ότι και τα μέλη τα αυτά τα τελευταία των Εθνικών Κοινοβουλίων έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεργαστεί με τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία εν ώψη και τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην κάθε χώρα μέλο, σε σχέση δηλαδή με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για του πολίτε τη. Ήδη η ΙΜΚΟ είχε διοργανώσει συναντήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εθνικό κοινοβούλιο σε σχέση με την οδηγία για τις καθυστερήσεις Πυρωμών και την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ σημαντική έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εσωτερική αγορά και χάρη σε μια θαυμάσια συζήτηση με τις χώρες μέλη, με την Κομισιόν, με το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να εκπονήσει ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, κάναμε μια συνάντηση για μια οδηγία που βρίσκεται συζήτηση όπου έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε μια οδηγία που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και βεβαίως θα έχουμε και τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην Εθνική Νομοθεσία, οπότε και για αυτό το θέμα θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέροντα και καρποφόρα θέματα για τα οποία θα έχουμε ενδιαφέρουσε συζητήσει. Σήμερα το απόγευμα, κατά τι 5.30-6 πατέρα, θα έρθει και ο, Ευρωπαϊ, ο Ευρωπαίο Επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ για τα θέματα που μα αφορούν. Ξέρετε ότι αύριο θα παρουσιάσει το Single Market Act, την πράξη της ενιαίας αγοράς στον τύπο Οπότε θα έχουμε αρκετές διαβουλεύσεις μαζί του και θα έχουμε αρκετή δουλειά. Δεν θα είναι συνέχεια μαζί μας βέβαια όλο το απόγευμα, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, διάθεσή του να συνεργαστεί μαζί μας για το θέμα που θα αντιμετωπίσουμε και θα συζητήσουμε σήμερα. Επίσης θα ήθελα βεβαίως να καλωσορίσω και τους εμπειρογνωμόνες που αποδέχτηκαν να έρθουν και να φέρουν τη δική τους προσωπική μαρτυρία για το τι έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων σε ευρω... Ε, προσόντων συγγνώμη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλωσορίζω λοιπόν τους κυρίους... Δεν ξέρω, ο κύριο Ιγουιτς Φούξ, δεν ξέρω αν είπα καλά το όνομά του, εκ μέρου ε, των Γερμανών Μηχανικών, ο κύριο Πατρίκ Φορτουή που εκπροσωπεί του φαρμακοποιού τη Γαλλία ο καθηγητής Τόνι Άζελ, πρόεδρος του Συμβουλίου Μεών και Νοσοκόμων Ηνωμένου Βασιλείου, η κυρία Μαρία Γκρος Πέτερσεν από τη Δανία, που εκπροσωπεί τη Δανία βεβαίως και παρουσιάζει το έγγραφο εργασίας που θα συζητηθεί αργότερα και που αφορά τέσσερα επαγγελμάτα. Στόχος λοιπόν της συνάντησής μας σήμερα είναι το να ακούσουμε τις απόψεις του κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου σε σχέση με την κατάσταση, με τα, διακυβευόμενα και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα των επαγγελματικών προσώπων, προσόντων συγγνώμη, και δεξιοτήτων. Ξέρετε όλοι ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση και γνωρίζουμε όλοι ότι η επαγγελματική επιτυχία διέρχεται από μια ανάγκη κινητικότητας, από κάποιες απαιτήσει μάλλον κινητικότητας, οι οποίες είναι πανευρωπαϊκές. Οπότε η συζήτηση αυτή αποτελεί μία από τις πρώτες συνεισφορές στην υποχρεωτική αναθεώρηση της οδηγίας εκ μέρους της Κομισιόν για τις επαγγελματικέ δεξιότητες, όπως θα σας πει και ο κύριος Μπαρνιέ στη συνέχεια, επειδή η Κομισιόν θα κάνει κάποιες αξιολογήσεις και μετά από τις αξιολογήσεις αυτές θα έχουμε μια πράσινη βίβλο το 2011 και θα ακολουθήσει βεβαίως και μια νομοθεσία για μια καλύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Γνωρίζετε επίσης ότι η πρόσφατη οδηγία του 2005 προκάλεσε πολλά προβλήματα μεταφοράς και πολλές χώρες ήταν κακοί μαθητές στη μεταφορά της οδηγίας, καθυστέρησαν πολύ για τη μεταφορά της οδηγίας αυτή όσον αφορά τις επαγγελματικέ δεξιότητες και προσόντα. Είχαμε μία αναγνώριση όλων των κοινών διπλωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 και μετά, κάτι το οποίο όμω δεν έγινε παντού, το οποίο σημαίνει θα πρέπει να επιταχύνουμε την προσπάθειά μας και θα πρέπει με τη βοήθεια των εθνικών αρχών να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην έχουμε τόσα προβλήματα και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται για τα θέματα αυτά επειδή όντως επίγουν. Η έκθεση της Κομισιόν για αυτή τη μεταφορά στην Εθνική Νομοθεσία της, της Οδηγίας του 2005 είναι διαθέσιμη και θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς και οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την ε, συλλογιστική ήδη παρουσίασαν κάποιες σκέψεις σε σχέση με την ουσία αυτής της οδηγίας. Δηλαδή έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την πολιτική, σε αυτή την ε, ομάδα εργασία από όλες τις πολιτικές ομάδες επειδή συνεργάστηκαν αρμονικά κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα εδώ στην Ευρωβουλή. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε αυτό το σύστημα και αυτό ακριβώς θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα. Δεν θα με ακρηγορήσω άλλο, απλά και μόνο για τους εκπροσώπου του εθνικών Κοινοβουλίου να πω ότι έχουμε κάποιους πολύ αυστηρούς κανόνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας δοθεί ο λόγος μετά τους εμπειρογνώμονες σε δύο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ακολουθήσει ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα ώστε όλοι, για να είναι όλοι μάλλον να, να είναι σε θέση να μιλήσουν θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε τρία λεπτά ομιλίας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμόρφωσή σας με αυτές τις απαιτήσει μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως τη συζήτησή μας και θα δώσω το, ρόλο, το λόγο στην κυρία Κάριν Μαρία Γκρός Πέτερσεν που θα μας παρουσιάσει αποτελέσματα του γράφου εργασία τη ΙΜΚΟ όσον αφορά τις δεξιότητε και τα προσόντα και που επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε τέσσερα επαγγελμάτα, νοσοκόμε, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ξεναγεί. Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω κάποιον από την Κομισιόν με τον οποίο συνεργάστηκα με μεγάλη χαρά και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Να, ευχα... να πάρα πολύ και να χαιρετήσω τον κύριο Τίτσα από την Κομισιόν επειδή θα πρέπει να το υπογραμμίσω δεν έχω ξανδει κάποιον που να εργάζεται τόσο καλά, να συνεργάζεται κανείς μαζί του τόσο καλά, να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα, με άμεσα τηλεφωνήματα, ας πούμε, και όχι με επιστολές που παίρνουν τρεις εβδομάδες. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και ελπίζω ότι μελλοντικά θα είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε και πάλι και ξέρω ότι έχετε συμμετάσχει ενεργά σε αυτό το φάκελο που έχει μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η κυρία Πέντερσαν έχει το λόγο. Okay. Thank you for the word, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα κάνω μία σύντομη παρουσίαση των βασικών πορισμάτων μιας πρόσφατης μελέτης ε, ε, εξ ονόματος Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Καταρχήν το ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής μελέτης και μετά τα βασικά ε, συμπεράσματα. Έξι συμπεράσματα διατυπώθηκαν μετά από τα πορίσματα. Ο στόχος της μελέτης ήταν η εξαγωγή ανάλυσης των προκλήσεων ε, για τέσσερα επελεγμένα επαγγέλματα διακινούμενων εργαζομένων όπου παρουσιάζονται προβλήματα, δηλαδή νοσοκόμοι, αρχιτέκτονες, πολιτική μηχανική και ξεναγή. Τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Δανία, Πολωνία, Σλοβενία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. 32 συνεντεύξεις από τα Εθνικά Σημεία Επαφής και τις Αρμόδιες Αρχές ε, καταγράφησαν και επίσης ε, από οργανώσεις, ενώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής μελέτης, από την αρχή αποφασίσαμε να αφιερώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις προκλήσεις που αναφέρονται. Στην χρήση της γραπτής δήλωσης εκ των προτέρων, περίοδος προσαρμογής ή επάρκεια, γλωσσικές προϋποθέσεις, συνεργασία και ρόλος των εθνικών ε, συνδέσμων και αρμοδίων αρχών, συστήματα εποπτείας και ανταλλαγή πληροφοριών για τον επαγγελματικό αποκλεισμό και την πληροφορία σχετικά με την επάρκεια, ε, επικύρωση επαλήθευση πληροφοριών για επαγγελματικά προσόντα, προστιθέμενη αξία μιας επαγγελματικής κάρτας και σχέσεις με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Επόμενο παρακαλώ. Πάμε στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη. Διαπιστώσαμε ότι οι επαγγελματίες έχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τις προσδοκίες τους γιατί δεν γνωρίζουν καλά την οδηγία και τις διαφορετικές, ε, τα, διαφορετικά χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν δυσκολίες να εντοπίσουν τις ομόλογες τους αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη-μέλη ε, αυτό το σύστημα ενημέρωσης εσωτερικής αγοράς, το IMI, ε, είναι καλό για τις αρμόδιες αρχές και θέλουν να χρησιμοποιείται ευρύτερα. Οι πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια ανταλλάσσεται ως μέρος της κανονικής διαδικασίας αναγνώρισης. Οι επαγγελματικές κάρτες μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία ε, αναγνώρισης, αλλά ακόμα υπάρχουν προκλήσεις σε σχέση με την εφαρμογή και ανάπτυξή τους. Επίσης, γραπτέ δηλώσει εκ των προτέρων χρησιμοποιούνται ω πρότυπο και βάση για τα περισσότερα κράτη-μέλη. Η αργή ενημέρωση του πέμπτου παρατήματο οδηγεί σε περισσότερες διαδικασίες αναγνώρισης με βάση το γενικό σύστημα που δημιουργεί μεγαλύτερο φόρτο. Τα μέτρα αντισταθμισή είναι πολύ απαιτητικά από άποψη πόρων και οι αρμόδιες αρχές δεν ξέρουν πώς θα αναπτύσσουν καλύτερα μέτρα. Η αναγνώριση είναι προβληματική εκεί όπου η πρόσβαση στο επάγγελμα δεν έχει ρυθμιστεί στο κράτος μέλος καταγωγής και τέλος η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προσόντα είναι χρονοβόρος και δύσκολη για τα επαγγέλματα στα πλαίσια του γενικού συστήματος αναγνώρισης. Όπως είπαμε, τα πορίσματα της μελέτης δείχνουν έξι συστάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις προκλήσεις για την αναγνώριση, ιδιαίτερα στα τέσσερα επαγγέλματα που, εξέτασαν, που εξετάστηκαν στη μελέτη. Η πρώτη σύσταση θα πρέπει η χρήση του IMI, του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς, να γίνει υποχρεωτικό και να ε, αναπτύξουμε, να το αναπτύξουμε περισσότερο. Η υποχρεωτική χρήση του IMI θα μειώσει τις καθυστερήσεις διαδικασίες αναγνώρισης και οι κανόνες που θα προσδιορίζουν ε, προθεσμίες για απαντήσεις θα μειώσουν τις ε, καθυστερήσεις. Πρόσθετα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι μια ενημέρωση ε, συναγερμού ή κατα... σημάτων για ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών για την επάρκεια και ένα σημείο επαφής διαλόγου για συζήτηση απαντήσεων που δόθηκαν σε ερωτήσεις. Η δεύτερη σύσταση είναι βελτίωση τη ενημέρωση του πέμπτου παρατήματο τη οδηγία. Αυτό στην πράξη, στην πράξη σημαίνει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν σε συχνά το παράρτημα. Επίσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν το παράρτημα στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας και με το ίδιο ε, τύπο πληροφοριών. Αυτό θα ε, οδηγούσε σε αποφυγή υπερβολικά σύνθετων προϋποθέσεων στο παράρτημα ή ε, παράληψη πληροφοριών. Αυτό θα μπορούσε να ε, γίνει μέσα από επικοδομητικό διάλογο μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την άλλη. Οι εθνικοί συντονιστές θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για τις εργασίες, αλλά θα πρέπει να στηρίζονται ενεργώς σε επίπεδο αρμόδιας αρχής. Η τρίτη σύσταση είναι να διασφαλιστεί αμοιβαία αναγνώριση, ακόμα και αν η πρόσβαση στο επάγγελμα δεν έχει ε, ρυθμιστεί στο κράτος μέλος καταγωγής. Αυτό στην πράξη μπορεί να γίνει ενισχύοντας το ρόλο των εθνικών σημείων επαφής στο κράτος μέλος καταγωγή σε σχέση με τα επαγγέλματα που δεν ρυθμίζονται. Επίσης, θα καθοδηγούνταν τα κράτη-μέλη σχετικά με το είδος της τεκμηρίωσης που συνιστά επαρκή απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων. Θα πρέπει όμως να υπογραμμιστεί ότι οι προσπάθειες για το μετριασμό αυτής της κατάστασης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε πιέσεις στα κράτη-μέλη που δεν ρυθμίζουν το επάγγελμα να αρχίζουν να το ρυθμίζουν. Τέταρτη ε, σύσταση. Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για διαδικασίες ε, που θα αναπτύσσουν μέτρα αντισταθμιστικά. Αυτό στην πράξη σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένα, βελτιωμένους τύπους αντισταθμιστικών μέτρων ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να συντονίζονται ειδικά εργαλεία. Μια πρακτική πλατφόρμα θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής ή η Ομάδα των Συντονιστών και επίσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές εφόσον εκείνοι γνωρίζουν τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει μέχρι τώρα. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε επίσης να υποστηρίζεται μέσα από την προαγωγή δικτύων για τις αρμόδιες αρχές για ιδιαίτερα ε, κινητικά επαγγέλματα, ε, για συζητήσει προβλημάτων ε, σε ατομική βάση και προσωπική. Πέμπτη σύσταση να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν προβλήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις σε σχέση με την τεκμηρίωση ε, διετούς εμπειρία σε περιπτώσεις γραπτής δήλωσης. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τη χρήση του άρθρου 7.2, ότι δηλαδή είναι μια προαιρετική διάταξη και μια απλή διοικητική διαδικασία Ενημέρωση, κοινοποίησης και όχι ένα πλήρως αναπτυγμένο σύστημα αδειών. Επίσης θα πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν κοινέ συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διμερός σχετικά με το τι ακριβώς θα σημαίνει και σε τι θα συνίσταται η απόδειξη της ε, πείρας ε, από την εργασία. Η τελευταία έκτη σύσταση είναι διευκόλυνση της ανάπτυξης των επαγγελματικών καρτών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει παρέχοντας γενικότερη υποστήριξη επικούρηση στην ανάπτυξη των ε, επαγγελματικών καρτών και βοηθώντας τις, τους οργανισμούς να μοιράζονται τη γνώση και την τεχνογνωσία πάνω στο θέμα. Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί ποια επαγγέλματα θα μπορέσουν να ωφεληθούν από μια τέτοια επαγγελματική κάρτα ή κάρτα του επαγγελματία και σας ευχαριστώ. Η πρόεδρος εκτός ναι, σημαντικό αυτό το, το έγγραφο και συγχαρητήρια που μειώσατε συγκεντρώσατε την παρουσίασή σας για να μην χάνουμε χρόνο στη συζήτηση. Το μεγαλύτερο τμήμα της συζήτησης θα επικεντρωθεί βεβαίως στην καταγραφή των αμοιβαίων επαγγελματικών αναγνωρίσεων και το δεύτερο τμήμα, αυτό το πρώτο και το δεύτερο τμήμα θα αφιερωθεί στις μελλοντικέ συστάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν για την αρμόνιση των επαγγελματικών προσόντων στην επικράτεια της Ένωσης. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ινξ Βίλι Φούτ, διευθυντή της Ομοσπονδίας Γερμανών Μηχανικών, που θα μας μιλήσουν για το τι γίνεται στον επαγγελματικό του τομέα στη χώρα του, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και για τις υπόλοιπες χώρες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Με παρακάλεσα να σας μιλήσω για τις γερμανικές εμπειρίες σχετικά με την διασυνοριακή αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μέσα από το πρίσμα των μηχανικών. Ευχαρίστως ανταποκρίνομαι στην παράκληση γιατί μπορώ να σας ενημερώσω όχι μόνο για τα γερμανικά πράγματα αλλά και για εκείνα των Ευρωπαίων μηχανικών. Έτσι, οι παρατηρήσεις μου αντικατοπτρίζουν τόσο τη θέση της Ένωσης των Γερμανών ε, Μηχανικών, VDI, της οποίας είμαι πρόεδρος, ε, όπως και τη θέση της Ομοσπονδίας των Ευρωπαίων, ε, Ευρωπαϊκών Ενώσεων Μηχανικών, ΦΕΑΝΗ. Καταρχήν, πολύ σύντομα, δύο λόγια για την Γερμανική Ένωση, ε, και τη ΦΕΑΝΗ. Το VDI είναι κοινοφελής οργάνωση με 139.000 μέλη, ε, είναι από, τους μεγα, τις μεγαλύτερες τεχνικές επιστημονικές ενώσεις της Ευρώπης, περίπου 130 πλήρους απασχόλησης μέλη, συντονίζουν την εργασία 13.000 εμπειρογνωμόνων που ε, προσφέρουν την τεχνογνωσία τους στην Ένωση και στους μηχανικούς. Με πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις, κατευθυντήριες γραμμές, μελέτες, γνωμοδοτήσεις, η Ένωση των Γερμανών Μηχανικών προάγει την επιστημονική ανταλλαγή και την κοινωνική συζήτηση για θέματα τεχνικά μεταξύ των ε, μηχανικών και των πολιτών. Η ΦΕΑΝΗ είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των ε, Μηχανικών εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ενώσεων των μηχανικών από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης συν ακόμα τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη. Ε, η Θεάνη μέσω των εθνικών οργανώσεων μελών εκπροσωπεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια μηχανικούς. Κυρίες μου και κύριοι, περνώ έτσι στο σημερινό μας θέμα. Οι επιχειρήσεις αλλά και οι παρέχοντες ε, υπηρεσίες μηχανικού, τα γραφεία μηχανικών ε, δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό στην Ευρώπη με την αυξανόμενη οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρώπη και για τους μηχανικούς η σημασία της διασυνοριακής κινητικότητας αυξάνεται. Η ανάγκη για διεθνώς διακινούμενους ε, ε, μηχανικούς στην Ευρώπη ε, αυξάνεται γιατί είναι διαφορετική η διαθεσιμότητα μηχανικών στις διάφορες χώρες. Η Γερμανία, για παράδειγμα, εδώ και χρόνια δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε ειδικού μηχανικούς και γερμανικές επιχειρήσεις ε, κάνουν ε, έντονες προσπάθειες να προσλάβουν από το εξωτερικό ειδικευμένους μηχανικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα εμπόδιο της κινητικότητας όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολες οι διαδικασίες για την διασυνοριακή αναγνώριση των προσόντων επαγγελματικών, ε, εκπαιδευτικών, μετεκπαιδευτικών. Στην Γερμανία η αρμοδιότητα για την αναγνώριση ε, βρίσκεται ανάλογα από το κρατήδιο είτε στην Προεδρία της Κυβέρνησης ή στη ε, επιμελητήρια των μηχανικών. Σε κάθε περίπτωση ε, υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να επικυρώνονται και να μεταφράζονται. Συχνά η διαδικασία κρατάει και έξι μήνες και στοιχίζει αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Σε άλλα κράτη-μέλη διαρκεί ακόμα περισσότερο αυτή η διαδικασία. Η Γερμανική Ένωση, η Ομοσπονδία Θεάνη, και τα, τα, οι οργανώσεις μέλη ε, θεωρούν ότι μια ταυτότητα επαγγελματική, μια κάρτα ε, επαγγελματική για τους μηχανικούς μπορεί να συμβάλλει στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Ήδη το 2005 η ΦΕΑΝΗ έκανε μια έρευνα σχετικά με τις ρυθμίσεις που υφίστανται στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών. Τη δημοσίευσε αυτή τη μελέτη. Και μετά η Γενική Συνέλευση του ΦΕΑΝΗ το Σεπτέμβριο του 2005 με βάση αυτή την έρευνα κατέληξε ότι θα πρέπει να αναπτύξει αυτή τη διαδικασία για την ταυτότητα και το 2010 τον Απρίλιο η Γερμανική Ένωση ε, κατέληξε στην απόφαση να επεξεργαστεί μια τέτοια κάρτα ή ταυτότητα και να την εφαρμόσει. Ε, το, συγγνώμη, το Σεπτέμβριο του 2005 έγινε αυτό και τον Απρίλιο του 2010 αποφάσισε η Γερμανική Ένωση ε, να ε, εισαγάγουν το, την επαγγελματική ταυτότητα για τους ε, μηχανικούς που λέγεται Engineering Card στη Γερμανία. Έγινε επιτυχώς αυτό. Η επεξεργασία έγινε σε στενή συνεργασία, η επεξεργασία έγινε σε συνεργασία με τα μέλη της ΦΕΑΝΗ. Στα πλαίσια των έντονων συζητήσεων διαπιστώθηκε ότι πέντε κριτήρια ε, είναι αποφασιστική σημασία για την αποδοχή και την επιτυχία αυτής της ταυτότητας. Πρέπει η ταυτότητα να είναι ε, ευρεία, τυποποιημένη, αξιόπιστη, αποκεντρωμένη και πέμπτον εθελοντική. Το τι σημαίνει αυτό λεπτομερώς θα σας το εξηγήσω. Ε, οι πληροφορίες ε, πάνω στην ταυτότητα η κάρτα είναι ε, ευρείες, δίνουν δηλαδή στοιχεία λεπτομερή για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. Δεύτερον, οι πληροφορίες είναι τυποποιημένες, διότι η engineering card αντικατοπτρίζει και παρουσιάζει πληροφορίες για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ε, για την ε, ακαδημαϊκή εκπαίδευση ισχύουν πάλι τα κριτήρια EURACE. Επίσης είναι αξιόπιστα τα στοιχεία πάνω στην ταυτότητα. Τα προσόντα ε, ελέγχονται και αναγνωρίζονται στη χώρα προέλευσης ε, από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία ε, αποτελείται από εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια, ενώσεις και την οικονομία. Έτσι διασφαλίζεται μια ευρία αναγνώριση της Engineering Card. Η παρακολούθηση της ε, Επιτροπής των Κρατών Μελών γίνεται μέσω της ΦΕΑΝΗ. Τέταρτον, η εισαγωγή και η διαχείριση της ταυτότητας της επαγγελματικής γίνεται αποκεντρωμένα σε επίπεδο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα αποκτηθέντα προσόντα στη χώρα προέλευσης, ε, τα προσόντα αυτά λοιπόν τεκμηριώνονται. Ε, πέρα από τις ε, τυποποιημένες καταγραφές ε, μπορούν να υπάρχουν και προσθήκες ανάλογα με το κράτος μέλος. Αυτή η ευελιξία για προσθήκες οφείλεται στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και στις ρυθμίσεις τις διαφορετικές ε, και προωθεί την αποδοχή των μελών θεάνη. Θα πρέπει να είναι εθελοντική, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να έχει την κάρτα αυτή κάθε μηχανικός ε, είναι μια υπηρεσία για τους μηχανικούς που θέλουν να είναι διεθνώς διακινούμενοι και έτσι διασφαλίζεται ότι η Engineering Card είναι μια λύση που ανταποκρίνεται σε ανάγκες και δεν ε, δημιουργεί επιπρόσθετες δαπάνες ή γραφειοκρατία. Ε, η Γερμανική Ένωση αλλά και η ΦΕΑΝΗ είναι πεπισμένη ότι η Engineering Card θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης. Τα μέλη ΦΕΑΝΗ ε, συμφωνούν λοιπόν και έτσι στη Γενική του Συνέλευση την 1η Οκτωβρίου του 2010 στη Σόφια ομόφωνα αποφάσισαν να ε, υιοθετήσουν την ε, engineering card και να την κάνουν κάρτα φεάνη οι ενώσεις των μηχανικών από 7 κράτη-μέλη είπαν ότι το 2011 θα την εισαγάγουν. Υπάρχουν και άλλα μέλη της ΦΕΑΝΗ τα οποία περιμένουν και την πολιτική υποστήριξη. Μια τέτοια υποστήριξη θα ήταν πολύ σημαντικό για την αναγνώριση. Μια τέτοια υποστήριξη ε, θα καθιστούσε την Engineering Card ως το κατεξοχήν όργανο για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ε, κινητικότητας των μηχανικών και θα ωφελούνταν και οι μηχανικοί στην Ευρώπη αλλά και οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις. Μια αντίστοιχη υποστήριξη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Engineering Card, ε, θα ήταν πάρα πολύ ευπρόσδεκτη και, για τη Φεάνη και ε, από τη ΦΕΑΝΗ και από το Γερμανική Ένωση. Σταματώ εδώ κυρίες και κύριοι και ε, περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Merci euh, Σας ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ήταν μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα συνθετική ε, εμπειρία. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βρίσκεστε εδώ σήμερα, έχετε λόγο που είστε εδώ, ε, μοιραζόμαστε όλοι τις ίδιες προσδοκίες και τις ίδιες ανησυχίες. Τώρα θα ανοίξουμε τη συζήτηση και θα ήθελα να πω στους βουλευτές και γερουσιαστές ότι είναι μεγάλη αίθουσα. Δεν βλέπω καλά τα καρτελάκια με τα ονόματα ε, για όσους θέλουν να πάρουν το λόγο, παρακαλώ, ε, υπάρχει αυτό το έντυπο το οποίο σας δείχνω τώρα. Ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν θέλετε να πάρετε το λόγο, να το συμπληρώσετε, έτσι ώστε να μην κατακρεουργήσω, λέει η Πρόεδρος, τα ονόματά σας, να ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει και παρότι αγαπώ πάρα πολύ τις γλώσσες δεν μιλάω πολλές. Λοιπόν, ε, θα έχουμε ε, εθνικούς βουλευτές και βουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τρία λεπτά ο καθένας, ανταλλαγή απόψεων. Τον, ρόλο, ε, τον λόγο συγγνώμη, έχει... Euh, η κυρία Γιούγκ, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι μέλος της Κοινωνικής Επιτροπής. Κυρία Γιούγκ, παρακαλώ. Baroness Jung. Και μάλιστα μπάρονες, Βαρόνι Γιούγκ θα έπρεπε να πω κανονικά. Σα Σας ευχαριστώ πραγματικά. Uh, Η οδηγία ε, την οποία γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ε, και την ε, οποία έχουμε μελετήσει την εποχή της σύνταξής της ε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Βέβαια το House of Lords δεν έχει ασχοληθεί ε, τελευταία με, την, ε, με το θέμα αυτό αλλά είχαμε την δυνατότητα να μελετήσουμε μία έκθεση από το House of Commons ε, η οποία αφορούσε το ίδιο θέμα. Βεβαίως, ε, ε, ειδικά στο ιατρικό επάγγελμα δημιουργούνται κάποια προβλήματα και έχουμε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την ανισότητα των, της κατάρτισης στις διάφορες χώρες. Πολύ πρόσφατα είχαμε τον θάνατο ενός Βρετανού, του κυρίου Ντέι, ο οποίος απεβίωσε μετά από μεγάλη μεγάλη δόση, υπερβολική δόση μορφήνης ε, που του χορήγησαν ε, στην Γερμανία από ένα Γερμανό γιατρό. Ε, δεν είναι δυνατόν εδώ βεβαίω δεν θέλω εγώ να αμφισβητήσω τις ικανότητες ενός γιατρού αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε έναν κατάλογο προσόντων που θα δίνεται και θα επιβεβαιώνεται από την πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας ε, σύμφωνα με τις ικανότητες ιατρικές και γλωσσικές που θα έχει ο γιατρός practitioner or otherwise to ensure their competence on the same. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, να έχουμε την ε, ίδια αντιμετώπιση, για προσόντα. Στην περίπτωση του θανάτου του κυρίου Ντέι, ο δόκτωρ Λουμπάνη ήταν βέβαια ήταν ικανός ιατρός αλλά προφανώς δεν είχε περάσει από ό,τι φάνηκε μετά τα τεστ γλωσσικής επάρκειας. All these matters Όλα τα θέματα αυτά συζητήθηκαν ε, κατά τη διάρκεια μιας διερευνητικής επιτροπής ε, του House of Law of Commons ε, και η επιτροπή είχε αποδεκτικά στοιχεία από πλευράς του GMC όπου θεωρείται ότι ότι η γλωσσική επάρκεια ήταν απαραίτητη ε, και, σύμφωνα με, ε, ε, με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αλλά από ό,τι κατά λέξη ανεφέρετο στην αναφορά τελικά είχαν λίγο χρυσώσει τη διαδικασία του 1993 και προφανώς έκαναν λίγο τα στραβά μάτια σε ορισμένες περιπτώσεις. Ε, το ε, GMC ε, ζήτησε νομική γνωμοδότηση και αποφάσισε ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να ζητήσει επισήμως από την κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερο αυστηρή όσον αφορά τις δοκιμασίες γλωσσικής επάρκειας αλλά και τις δοκιμασίες επαγγελματικής ικανότητας. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι αρμόδιες αρχές να συνεργάζονται έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, οποιαδήποτε αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει οπωσδήποτε ε, και πρόκειται να μελετάτε ενδελεχώς από την European Scrutiny Committee του House of Lords και του House of Commons πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, μελετήσουμε προσεκτικά ε, και ε, τις, εξετάσεις γλώσσας οι οποίες αναφέρονται στις κλινικές δοκιμές η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών όπως άλλωστε προβλέπεται από την ε, υφιστάμενη οδηγία δεν λαμβάνει η χώρα σε ικανοποιητικό βαθμό. Ναι, ναι, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε. Ε, γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου επαγγελματίες οι για τους οποίους έχει απαγορευτεί ε, η άσκηση του επαγγέλματός του σε μια χώρα εξακολουθούν να είναι σε θέση και να έχουν την ικανότητα να ασκούν το ίδιο επάγγελμα σε μια άλλη χώρα. Ε, επομένως όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και να μελετηθούν εμβριθώς για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή. Ευχαριστώ για την μαρτυρία σας. Θα το συζητήσουμε στο δεύτερο τμήμα για την ασφάλεια των ασθενών και την ασφάλεια για των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Μιλήσαμε για την εσωτερική αγορά, αναφερθήκαμε στο σύστημα ΙΜΗ και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους από την Ιταλία, από τη Βουλή της Ιταλίας, ο κ. Σινιάτσο Αμπριάνη. Η Νιάτσο Βρυγιάννη από την ε, Βουλή και εξ ονόματος ε, του συνόλου του σώματος σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκλησή σας. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων βεβαίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν μεγάλο τμήμα του τριτογενούς τομέα και αυτό καταδεικνύει τα λεγόμενά μου ακόμα περισσότερο. Από τη μία πλευρά ε, η επιτάχυνση και η βελτίωση των διαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ε, μπορεί να ε, προωθήσει υπέρ των καταναλωτών την αναγνώριση των εν λόγω προσόντων. Επίσης να δημιουργήσει καλύτερες και πλέον κατάλληλες οικονομικές συνθήκες. Μας εκπλήσει βεβαίως το γεγονός ότι μονάχα για 7 επαγγελματά από τα 80 και τόσα που ε, υπάρχουν στην Ευρώπη αναγνωρισμένα, υπάρχει αυτή ε, η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Άρα πολλά μπορούν ακόμα να γίνουν, πολλές βελτιώσεις μπορούν ε, να υπάρξουν. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αναγνώρισης να μπουν σε αυτό το σύστημα φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο η διασφάλιση ε, των πολιτιστικών ε, συνθήκων και να μην υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είτε πρόκειται για δικαίωμα στην περίθαλψη είτε πρόκειται για θέματα άμυνας πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν δικαίωμα, ε, στην, ε, έχουν δικαίωμα σε υψηλής ποιότητος ε, υπηρεσίες. Ε, στην Ιταλία έχουμε πολλές φορές ε, περιπτώσεις ε, ανθρώπων οι οποίοι έρχονται με διπλώματα από σχολές φαντάσματα, από πανεπιστήμια φαντάσματα και που παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα να επιβεβαιώσουν τους τίτλους τους και να αναγνωρίσουν τους τίτλους σπουδών τους. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Ε, στην χώρα μου την Ιταλία οι ιδεοντολογικές ε, αρχές ε, καταγράφονται σαφώς βάσει συγκεκριμένου νόμου. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή μελετάει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του συνολικού θέματος και ο υποφαινόμενος είναι εισηγητής για τη μεταρρύθμιση αυτή. Οι ε, οργανώσεις επίσης των, ε, οι οργανώσεις των ε, επαγγελματιών είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να μας βοηθήσουν. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κάθε φορά για να ακούμε προσεκτικά τι λένε και οι επαγγελματίες. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε ακριβείς στο χρόνο σας, αλλά δυστυχώς, λέει η Πρόεδρος, προκαλέσετε κάποια προβλήματα στους Γερμηνείς γιατί πηγαίνατε πάρα πολύ γρήγορα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο, σε ένα μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην κυρία Ευλίν Γκέμπαρτ. Είναι συντονίστρια λοιπόν τη σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε ο Ιταλός συνάδελφος. Ήδη δηλαδή μπορούμε να συναγάγουμε ένα συμπέρασμα σήμερα ότι το σύστημα ήμι πρέπει να βελτιωθεί. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον έλεγχο αν είναι γνήσιο ή όχι ένα υποβαλλόμενο πτυχίο μέσα από αυτό το σύστημα το σύστημα πληροφόρησης ή ενημέρωσης ε, εσωτερικής αγοράς, το ΙΜΗ. Ερωτήσεις τώρα. Μία ερώτηση στην κυρία Πέτερσεν. Πρόκειται για το εξή ερώτημα. Η περίοδος προσαρμογής ή η επάρκεια, το τεστ επάρκειας. Τότε με την οδηγία έγινε μεγάλος καυγάς μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ποιος θα αποφασίζει δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Το τεστ, η εξέταση, ε, ο διαγωνισμός καθ' αυτός ή μια περίοδος προσαρμογής. Και εμείς είπαμε ότι ο ίδιος ο υποψήφιος δύο θα το αποφασίζει αυτό. Γίνεται όμως αυτό. Θα με ενδιαφέρει να το ξέρω τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Και σε αυτά τα πλαίσια, κοιτάζοντας τον κλάδο των ξεναγών, παρατηρώ ότι πολλές τέτοιες εξετάσεις και περίοδοι υπάρχουν σε ένα κράτος μέλος, στην Ιταλία συγκεκριμένα. Το έχουμε εξετάσει να το δούμε. Γιατί δηλαδή στο ένα κράτος γίνονται πολύ περισσότερα τέτοια πράγματα από ότι σε κάποια άλλα. Τι κρύβεται από πίσω. Θα με ενδιαφέρε. Ερώτηση προς τον κύριο Φούξ. Να σας το ξεκαθαρίσω εξ ονόματος της ομάδας μου, της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας, ότι αυτή την επαγγελματική ταυτότητα η κάρτα σίγουρα την υποστηρίζουμε. Αυτό μεταξύ άλλων εμείς το υποβάλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι πρόκειται για ε, ένα μη συμβατικό μέσον, μη γραφειοκρατικό μέσον για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα διακινούνται στην Ευρώπη και είναι καλό πράγμα αυτό. Συμπληρωματική ερώτηση. Τώρα λέτε ότι θεσμοθετήθηκε. Υπάρχουν πλέον μηχανικοί που την έβγαλαν την κάρτα και πού είναι. Πόσοι μηχανικοί έχουν βγάλει την κάρτα αυτή. Η ζήτηση είναι πραγματικά μεγάλη για αυτή την κάρτα. Είναι κάτι που εμείς το βρίσκουμε θεωρητικά και από μακριά ωραία, ενώ δεν λειτουργεί στην πράξη. Πολύ θα με ενδιαφέρε να μου το πείτε αυτό. Πριν να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις, για να μην ξεφύγουμε από το πνεύμα των ερωτημάτων που τέθηκα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πίτεσαν και στον κύριο Φούξ για να απαντήσουν στα σημαντικά ερωτήματα της κυρίας ε, Γκέπαρτ. Κυρία Πίτερσεν. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω μόνο δύο λόγια. δεν είχαμε δυνατότητα να πάμε σε μεγάλο βάθος λεπτομέρειας. Γι' αυτό ακριβώς κοιτάξαμε το ότι υπάρχει και το ότι χρησιμοποιείται στις χώρες μέλη. Όσον αφορά λοιπόν τις, τους οδηγούς και τους... Ε, συγγνώμη. Αυτά τα επαγγέλματα και τους χρόνους προσαρμογής και τις μεταβατικές περιόδους για τους ξεναγούς ας πούμε. Κοιτάξαμε τι γίνεται στις διάφορες χώρες αλλά επειδή ακριβώ ε, Ξαναλέω, δεν είχαμε πάει σε λεπτομέρειες επίπεδο ανάλυσης, δεν ε, αναφέραμε ε, συγκεκριμένα παραδείγματα και στοιχεία, απλά και μόνο κοιτάξαμε τι είχαμε διαθέσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκέμπχαρτ, Ευχαριστούμε καταρχήν πολύ για την υποστήριξη. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά για την επαγγελματική ταυτότητα η κάρτα. Τον Απρίλιο στην έκθεση του Ανοβέρου πρώτη φορά παρουσιάσαμε αυτή την κάρτα για τη Γερμανία και μπορούμε να πούμε ότι μέχρι σήμερα περίπου 200 κάρτες έχουν ήδη δοθεί. Το δεύτερο σημαντικό βήμα έγινε στη Σόφια την 1η Οκτωβρίου όπου ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της ΦΕΑΝΗ ε, ψήφισε υπέρ της κάρτας και όλοι θα την προβάλλουν. Εμείς ε, το θέλαμε αυτό. Το τρίτο βήμα είναι να γίνει επίσημο έγγραφο. Οπότε θα ακολουθήσουν και όλες οι άλλες χώρες. Είπα, ε, τα χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάρτα. Ε, η επόμενη χώρα θα την εισαγάγει, θα είναι η Ολλανδία. Και θα αρχίσει να την βγάζει, να την εκδίδει στις αρχές του επομένου έτους. Μέχρι το τέλος του επομένου έτους ο στόχος είναι να έχει μπει η κάρτα τουλάχιστον σε 10 ευρωπαϊκά κράτη. Και έτσι... Ε, θα αυξηθεί και η ζήτηση. Πολλές γερμανικές επιχειρήσεις ήδη, κυρίως μικρομεσαίες, μας ενημερώνουν ότι αυτή η κάρτα είναι μεγάλο βοήθημα. Γιατί μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζομένους από όλη την Ευρώπη, αλλά στις μικρές επιχειρήσεις δεν ξέρουν, δεν μπορούν να ξέρουν αν όντως ο υποψήφιος είναι ή δεν είναι μηχανικός. Γι' αυτό η γερμανική οικονομία μας υποστηρίζει εδώ εμπράκτος και στεναρός. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι απαντήσεις ήταν ε, ξεκάθαρες. Θα δώσω τότε το λόγο τώρα στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιταλικής Ιερουσίας, την κυρία Ροζάνα Μπόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την αυτονομή αναγνώριση των διπλωμάτων και συγκεκριμένα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Οδοντίατροι. Ιταλοί με πτυχίο ρουμανικό και με αίτηση στο αντίστοιχο δικατσά για αναγνώριση. Αυτοί οι πολίτες δεν πάνε σε κανένα μάθημα, δεν κάνουν τίποτα. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που οι Ιταλικές αρχές ξεκίνησαν μια ποινική διαδικασία όπως επίσης και οι Ρουμανικές αρχές. Η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε διμερή συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή της Ρουμανικής κυβέρνησης αλλά δεν έχει συμβεί ακόμα τίποτα και θα έπρεπε να ζητήσουμε μια πιο στενή συνεργασία των αρμόδιων αρχών των χωρών μελών γενικά για τέτοιου είδους προβλήματα. Επίσης υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την πιστοποίηση κατάρτισης ή διπλωμάτων που προέρχονται από κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επειδή αυτές οι χώρες πιστοποιούν ως συγκρίσιμα ή αντίστοιχα μαθήματα διάρκειας ενός έτους που σε άλλες χώρες κρατούν τρία χρόνια. Δεν αναφέρεται δηλαδή ξεκάθαρα το μάθημα στο οποίο φίτησε κανείς. Οπότε θα ήταν καλό και αυτό να το εξετάσουμε περισσότερο εις βάθος. Επίσης, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έχουν λάβει κοινοτικοί πολίτες σε τρίτη χώρα αναγνωρισμένοι από τη χώρα μέλος και πάλι οι αρμόδιες αρχές και στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο Υγείας αλλά και άλλες αρχές εξετάζουν πολλές περιπτώσεις ε, διπλωμάτων που λύθηκαν στην Σερβία και στο Μακρο, Μαυροβούνιο που αναγνωρίζονται στην ε, Ρουμανία και που μετά πήγαν στην Ιταλία. Είχαμε κάποια αντίδραση από τις Ιταλικές αρχές, παρόλα αυτά όμως οι Ρουμανικές αρχές συνεχίζουν να γνωρίζουν αυτά τα διπλώματα και πολλές φορές είναι διπλώματα από ανύπρακτα πανεπιστήμια όπως το Capital University που πραγματικά δεν υπάρχει. Επίσης θα ήθελα Α, ολοκληρώνω πρόεδρε γιατί βλέπω ότι τέλειωσε ο χρόνος μου. Τέλειωσα. Τέλειωσα. Ευχαριστώ. Α, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν δικός μου χρόνος. Διάβασα το τρία. Να προσθέσω λοιπόν σύντομα. Λυπάμαι, πρόεδρε. Λυπάμαι, πρόεδρε. Κοιτάξτε, να πείτε δύο λογάκια, πείτε τα. Ευχαριστώ. Το Εθνικό Συμβούλιο Ιταλών Μηχανικών μας αναφέρει ότι οι Ιταλοί πολίτες οι οποίοι έχουν κατάρτιση βιομηχανικού εμπειρογνώμονα πηγαίνουν στην Αγγλία για να εγγραφούν σε ένα οργανισμό επαγγελματικό και να λάβουν το πτυχίο του μηχανικού. Μετά γυρνούν στην Ιταλία και θεωρούν ότι έχει αναγνωριστεί το δίπλωμα του μηχανικού. Βεβαίω, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θέλω να επισέλθω στο αγγλικό σύστημα ή να κριτικάρω το αγγλικό σύστημα παροχή διπλωμάτων, αλλά βεβαίω εδώ πρόκειται ξεκάθαρα για μια περίπτωση παράκαμψη τη αλληλική ε, νομοθεσία, το οποίο σημαίνει βεβαίω ότι η οδηγία που αναφέραμε προηγουμένω το 2005 παρουσιάζει κάποια παράθυρα και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Πρόεδρο. Θέσατε κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα που νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκαν και στην ομιλία του κυρίου Φούξ εγώ σημείωσα ότι αυτά τα διπλώματα θα πρέπει να είναι αντικείμενο πολίθευσης από μια ανεξάρτητη αρχή με εμπειρογνώμονες κτλ. Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν, να, να ήταν μια λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζεται στην Ιταλία. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Νομίζω ότι ένας μόνο από τα εθνικά κοινοβούλια ε, θέλει το λόγο. Οπότε κοιτάξτε, ε, ξαναλέω, έχετε αυτό το χαρτί να σημειώσετε το όνομά σας αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Ο κ. Φεσνέρ, που είναι μέλος τη Επιτροπή για την Αγνώριση των Επαγγελματικών Διπλωμάτων και ο οποίο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και μάλιστα τότε ήταν ένα ευρύτατο και δύσκολο θέμα που μας απασχόλησε. Είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη που έγινε. Δεν θέλουμε να δούμε τις εκατοντάδες παράπονα μεμονωμένα που φτάνουν μέχρι εμάς τους βουλευτές, αλλά να καταλήξουμε σε κάποιες δομές και να προχωρήσουμε ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμένα. Ο δόκτωρο Φούξε μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Η μηχανική είναι πολύ καλά οργανωμένη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάτε μια κοινή γλώσσα μηχανικών μάλιστα ναι. πλέον, γιατί υπάρχουν πλατφόρμες που διευκολύνουν τα πράγματα, ενώ σε άλλους τομείς οι διαφορές είναι μεγάλες. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που ρυθμίζονται σε κάποιες χώρες, σε άλλα όχι. Και είναι δυσκολία ο συνδυασμός και η συνεννόηση. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ε, από τη δική σας περίπτωση, τι γενικότερα συμπεράσματα μπορούμε να ε, συναγάγουμε. Επίσης, θα έκανα μια διαφοροποίηση μεταξύ δύο περιπτώσεων. Αν κάποιος, ας πούμε, προσωρινά πάει να παράσχει υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος ή εάν θα εγκατασταθεί μόνιμα εκεί και θα απασχοληθεί σε κάποιο γραφείο μηχανικών. Γίνονται διαφοροποίησεις μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Είναι δυνατόν να γίνει κάποια διαφοροποίηση ή θα αντιμετωπιστούν και οι δύο περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι ερώτηση και στους δυο σας. Δηλαδή, μόνιμη εγκατάσταση σε κάποιο κράτος μέλος αν αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το αν κάποιος προσωρινά ε, παράσχει μια υπηρεσία σε ένα άλλο κράτος μέλος. Υπάρχουν διαφορές ό,τι αφορά την ε, άδεια που θα δοθεί ή γίνεται κάτι τέτοιο. Διαφοροποιημένη προσέγγιση. Euh, Κύριε Λέσνερ, θέσατε ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί είναι αλήθεια ότι η προσωρινή κινητικότητα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ουσιώδες αυτό το ερώτημα και πρέπει να το θέσουμε. <clears throat> Είναι σημαντικό το θέμα ε, να υπάρχει ασφάλεια. Είτε, δηλαδή να εργάζεται και να προσφέρει ασφάλεια ο μηχανικός, είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Τώρα, αν μπορεί κανείς να συναγάγει γενικότερα συμπεράσματα από τους μηχανικούς. Χαίρομαι που μας θεωρείτε έτσι καλά οργανωμένους. Το θέμα της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης το λύσαμε εμείς με μια διπλή διαδικασία σε δύο επίπεδα. Πρώτον, είναι σημαντικό οι σπουδές να ε, πιστοποιηθούν με βάση τα ευρωπαϊκά ε, πρότυπα πιστοποίησης και να είναι διαπιστευμένος ο φορέας της αναγνώρισης. Αλλιώς ο πτυχιούχος δεν μπορεί να πάρει την άδεια εκτός και εάν αποδείξει ε, ισοδυναμία με τα κριτήρια de juris. Και επίσης υπάρχει και μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία μπορεί επίσης να αξιολογήσει το σύστημα και είναι από μέλη που είναι στο Μητρό και επίσης γίνεται ε, συνεχής παρακολούθηση μέσα από την Ομοσπονδία Θεάνη γιατί υπάρχουν και απόπειρε χειραγώγηση του συστήματος. Αλλά εμείς έχουμε ένα ε, ε, σύστημα τριών επιπέδων που μπορεί να το μιμηθούν και άλλα επαγγέλματα και έτσι ε, ελαχιστοποιούμε, γιατί δεν μπορεί κανένα σύστημα να αποκλείσει τέτοιου είδους ε, παρατράγουδα, αλλά τουλάχιστον τα ελαχιστοποιούμε. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Φρανσίς Αζιούς, εκ μέρους του Κοινοβουλίου της Μάλτας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφέρατε πολύ σωστά το όνομά μου κατάγομαι από την μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι πολύ που σήμερα τα Εθνικά Κοινοβούλια λαμβάνουν το λόγο σε ένα διεθνές φόρουμ. Εγώ είμαι γιατρός αλλά είμαι και ακαδημαϊκός διδάσκος στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Μάλτα που έχει μόνο ένα πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές είναι μεσαίου μεγέθους και είναι σημαντικό για μας να αναγνωρίζονται τα πτυχία μας, όχι μόνο για τους φοιτητές μας, αλλά και για τις ευκαιρίες απασχόλησης, για την ίδια την κινητικότητα, λόγω ελλείψεως κάποιων μαθημάτων ή ειδικεύσεων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ενδεχομένω στον τομέα της τεχνολογίας, τη επιστήμης κλπ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και για τους φοιτητές μας το θέμα αυτό. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό και για αυτού που θα θέλαν να έρθουν να εργαστούν στη χώρα μας. Έχουμε πολύ καλή νομοθεσία σε πολλούς τομεί Έχουμε και σώματα όπως το Ιατρικό Συμβούλιο το οποίο ρυθμίζει την, τον τομέα των νοσοκόμων και θα ήθελα να πω ότι τα επαγγέλματα αυτά προστατεύονται, ρυθμίζονται σωστά. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με την εναρμόνιση. Αν κάποιος λοιπόν αποφασίσει να γίνει νοσοκόμος, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλα κενά και διαφορές μεταξύ ας πούμε Μάλτας και Σλοβενίας. Από ό,τι είδαμε όμως υπάρχουν διαφορές, επειδή υπάρχουν κάποια ιδρύματα ακαδημαϊκά, τα οποία δεν υπάρχουν ανύπαρκτα ή δεν είναι ιδρύματα ακαδημαϊκά. Πολλές φορές βεβαίως αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, αποτελεί μια αυθαιρεσία και δημιουργεί μεγάλα σοβαρά προβλήματα, επειδή κάποιος λαμβάνει ένα πτυχίο ή ένα δίπλωμα το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει. Εκεί λοιπόν αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια κατάσταση η οποία θα βλάψει όχι μόνο αυτό που λαμβάνει το δίπτωμα ή το πτυχίο αλλά και άλλους πολίτες. Ο κ. Φόξ ας πούμε είναι μηχανικός, δηλαδή ένας τομέας για τον οποίο δεν έχω μεγάλη γνώση. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί μηχανολόγοι, υπάρχουν χημικοί μηχανολόγοι, υπάρχουν ε, πολιτικοί μηχανικοί. Ε, εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε για τα άτομα που ψάχνουν δουλειά να έχουν καλώς καθορισμένα προσόντα για να βρουν καλύτερα και πιο εύκολα δουλειά και για να ευκολούν δηλαδή τους πιθανούς εργοδότες τους να τους εντοπίσουν Υπάρχουν τομείς σήμερα οι οποίοι εξελίσσονται όπως τεχνολογία, όπως και άλλοι τομείς και που έχουν να κάνουν και με την ιατρική, οι ορθοδοντικές που στο κόμες, οι δοντίατροι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τομείς συγκεκριμένα να έχουμε μια πλήρη νομοθεσία. Επίσης να πω ότι η χώρα μας ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ε, Μπολόνια, της συνθήκης και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το θέμα της εναρμόνισης των σπουδών. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να κινηθούν εύκολα από μια χώρα στην άλλη και να έχουν πρόσβαση όλοι στην γνώση εξίσου. Θα έπρεπε λοιπόν να διευκολυνθούν στη συνέχιση των σπουδών τους, θα πρέπει εμείς να τους παράσχουμε αυτή τη δυνατότητα να τους διευκολύνουμε όσο μπορούμε, να αυξήσουμε την κινητικότητά τους και να πω επίσης, τελειώνοντας, δύο λόγια για τα μαθήματα στο ίντερνετ ή τη φίτηση μέσω ίντερνετ που αυξάνεται διαρκώς. Δεν θα πω μ, κάτι το αρνητικό ενδεχομένως, δεν θα κάνω κάποια κριτική αρνητική, αλλά βλέπω ότι αυτά τα μαθήματα μέσω ίντερνετ αυξάνονται συνεχώς, ε, ρυθμίζονται, αλλά νομίζω θα πρέπει να τα κοιτάξουμε λεπτομερέστα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σημεία τα οποία αναφέρατε και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η κινητικότητα των νέων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ουσιώδου σημασία για την επιτυχία που θα έχουν στο επαγγελματικό τους ε, μέλλον. Μιλάμε για τον έρασμο και μετά δημιουργήσαμε ε, και τον ε, έρασμους για μαθητευόμενους, για μικρές επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν και όλες αυτές οι μελέτες στις οποίες αναφέρεται. Είδαμε, είδαμε επίσης τα όρια του, της διαδικασίας της Μπολόνιας. Κύριε Φούς, φαίνεται ότι όλοι εσάς θέλουν να απαντήσετε, όλοι σε εσάς κάνουν ερωτήσεις. Μια και σας έχουμε λοιπόν εδώ και έχουμε και λίγο χρόνο, Απαντήστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι η engineering card πρέπει να ειδωθεί ε, μόνο πρώτον σε σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνια και δεύτερον με τη σχετική διαδικασία διαπίστευσης, δηλαδή τα πρότυπα ποιότητας. Είπατε από πού θα καταλάβω ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι σε θέση να κάνει τη δουλειά για την οποία το θέλουμε. Πέρα από τα, το αν θα είναι πολιτική, μηχανική, ηλεκτρολόγη, μηχανική ή οτιδήποτε, οι σπουδές είναι διαρθρωμένες έτσι ώστε να υπάρχει ένα ε, διπλώμα supplement, ε, συμπληρωματικές σπουδές, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια. Και έτσι φαίνεται ποια μαθήματα παρακολούθησαν και με ποια επιτυχία ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα μαθήματα αυτά. Έτσι λοιπόν ένας τρίτος μπορεί αμέσως να ξέρει ποια προσόντα ακριβώς διαθέτει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεύτερον, είναι σημαντικό και εμείς ως θεάνοι το ζητήσαμε ρητά αυτό, αυτές οι εκπαιδευτικές κλίμακες να ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα. Και αυτό ε, αυτά τα, προ... τα πρότυπα τα αναπτύξαμε και είναι τα γνωστά πρότυπα ε, de jures. Πρέπει λοιπόν να συμφωνούν με τη διαδικασία της Μπολόνια και δεύτερον να έχει περάσει από το γιούρες η απίστευση. Αυτό είναι μια σφραγίδα ποιότητας και μπορεί κανείς να είναι ε, σε μεγάλο βαθμό βέβαιος ότι αυτά που αναφέρονται στο πτυχίο ε, τα καλύπτει ο υποψήφιο ο μηχανικός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση για την αποδοχή ε, μιας τέτοιας επαγγελματικής ταυτότητας. Εδώ δείξαμε μεγάλη συνέπεια. Κινηθήκαμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και όλα αυτά από κοινού κάνουν το σύστημα, θεωρούμε, απόλυτα πρακτικό, με ελάχιστη, ελάχιστα γραφειοκρατικό, ε, πολύ διαφανές και ε, αποτελεσματικό. Ε, la Το λόγο έχει ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων είναι βασική αρχή της εσωτερικής αγοράς και Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρξει καλή κινητικότητα, ε, συγγνώμη, δεν, δεν μπορεί να υπάρξει καλή κινητικότητα εάν ε, κάποιο δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του σε μια άλλη χώρα. Ε, Βεβαίω συμφωνούμε με την επαγγελματική κάρτα και μπορεί να αποτελέσει καλό εργαλείο για κάθε επαγγελματία που θέλει να εργαστεί σε μια άλλη χώρα. Από την άλλη πλευρά, βεβαίω θα πρέπει να δούμε από πάρα πολύ κοντά την τεχνική βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος ε, γιατί είναι δύσκολο. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι πληροφορίες να είναι σωστές, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες θα μπαίνουν ε, σε αυτήν την κάρτα. Μην ξεχνάτε όλες τις δεσμεύσεις και περιορισμούς που έχουμε ε, λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επομένως θα πρέπει να δούμε πόσος δρόμος μας χωρίζει από την κάρτα αυτή. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και διοικητική συνεργασία. Θα ήθελα επίσης γνώμη της κυρίας Πέτερσον όσον αφορά αυτήν την πρώτερη δήλωση. Γιατί δεν είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο από όλους τους επαγγελματίες όπως φαίνεται να υπονοούν τα κράτη-μέλη. Ε, κατά την άποψή μου ε, η ευρεία εφαρμογή αυτής της αρχής ενδεχομένως θα αποτελέσει εμπόδιο ε, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εάν απαιτείται και είναι προϋπόθεση για όλους τις επαγγελματίες. Νομίζω ότι μια καλή λύση θα ήταν οι αρμόδιες αρχές ε, να αποφασίσουν αν χρειάζεται πρώιμη ή πρώτερη δήλωση ή εν πάση περιπτώσει πρώτερη ε, εγγραφή σε κάποιο μητρό. Ε, θέλουμε επομένως να έχει η εθνική διοίκηση δυνατότητα διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά στο θέμα αυτό και εν περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει αναπερίπτωση ε, επίσης να πω στην συνάδελφο από την Ιταλία ότι δεν ξέρω κανέναν ε, που να ε, στη χώρα μου είτε είναι Ρουμάνος είτε είναι Ιταλός που να μην έχει τέτοιο κανονικό πτυχίο από Ρουμανικό Πανεπιστήμιο. Ακούγοντας αυτά πραγματικά μένω έκπληκτος και οπωσδήποτε θα έρθω σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές της χώρας μου έτσι ώστε να λάβω όσο γίνεται περισσότερες εξηγήσεις για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Στάιλερ, παρακαλώ. Κάθριν Στάιλερ, ναι. Από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω, κυρία Πρόεδρε. Μερικές σύντομες ερωτήσεις και σε σχέση και με αυτό που είπε και η Βαρόνι Γιάνγκ προηγουμένως Ενδεχομένως μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω σχετικά με το πώς ε, φέρνετε σε επαφή όλους τους κλάδους των μηχανικών, γιατί αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Επίσης, ποιο είναι το κόστος της ε, κάρτας. Επίσης, ε, αναπτύσσεται κάποιο τρόπο μέσω του οποίου ε, μπορείτε να ελέγξετε ε, επιγραμμικά online ε, τις διάφορες τα διάφορα προσόντα, δηλαδή φαίνονται online, εμφανίζονται online όλα αυτά τα προσόντα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην προκείμενη περίπτωση την ηλεκτρονική επικοινωνία και σε σχέση με αυτά που είπε η Βαρόνι Γιάνγκ, βεβαίως μας ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας στην παροχή των ε, υπηρεσιών ε, υγείας, ειδικά για, ε, για το επάγγελμα το ιατρικό, θεωρούμε ότι βεβαίως ε, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ε, έχουμε και την αναγνώριση ε, των παραγιατρικών επαγγελμάτων μέσω της δηλώσεως του Βερολίνου. Βερολίνου. Η Βαρονή αναφέρθηκε στο παράδειγμα του κυρίου Λουμπάνη, αλλά νομίζω ότι και στην Ισπανία πρόσφατα υπήρχε ένας γιατρός από την Αργεντινή, ο οποίος είχε διαγραφεί από ε, από τον Ιατρικό Σύλλογο στην Ισπανία και που όμως παρόλα αυτά μπόρεσε να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και να ε, ασκήσει το επάγγελμά του. Ε, νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να δούμε λίγο αυτά τα πράγματα και ακούμε εδώ πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και ο κύριος Μπουζόη αυτό που είπε η Ιταλίδα συνάδελφος πρώτη φορά το άκουγε για την ύπαρξη αυτού του πανεπιστημίου είναι καλό λοιπόν που μας ανοίγετε εδώ τα μάτια θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ και μετά η κυρία Πέιτερσεν ενδεχομένως ε, γιατί ε, δεχτήκατε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την πρώτερη δήλωση, είχατε και τις ε, ερωτήσεις της κυρίας Στάιλερ. Η Μπάρμπαρα Βάιλερ και μετά η κυρία Πέτερσεν για να απαντήσει. Δύο ερωτήσεις. Είμαι μεταξύ των συναδέλφων που με μεγάλο ενθουσιασμό και ζήλο ε, συνέβαλαν στην ε, έγκριση της οδηγίας, την υιοθέτησή της, νέβη καταφατικά η συνάδελφος από τους πράσινους, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν πολύ θετική και ίσως ό,τι την αύξηση των διακινουμένων εργαζομένων, αλλά, και το λέω κάπως ε, επικριτικά, και αυτό αφορά τη Γερμανία, ε, ε, σπάει μια στενοκεφαλιά που υπάρχει. Ότι δηλαδή κάθε χώρα πιστεύει ότι έχει τους καλύτερους μηχανικούς. Καταρρύπτονται αυτά τα ταμπού και τα, οι προκαταλήψεις. Ε, ξεναγή μπορεί να μην είναι ρυθμισμένο επάγγελμα στη Γερμανία. Στην Ιταλία μπορεί να είναι. Και υπάρχουν δυσκολίες οι Γερμανοί και άλλοι Σκανδιναβοί, για παράδειγμα, να ε, ε, εργάζονται σε κάποιες χώρες. Εξακολουθεί να είναι κλειστό το επάγγελμα σε κάποια επαγγέλματα σε ορισμένες χώρες ή συμβάλλουν όλα αυτά στο άνοιγμα της αγοράς. Δόκτωρ Φούξ, νομίζω ότι αυτά που μας είπατε είναι το καλύτερο που μπορεί κανείς να φανταστεί είναι οι μέγιστες προσδοκίες μας. Σε... Θυμάμαι μια ακρόαση που ρωτήσαμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο γιατί χρειάζονται τόσες διαδικασίες και γιατί δεν εφαρμόζεται σωστά η οδηγία. Και μας είπαν ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αφενός, αλλά αφετέρου υπάρχουν και αντιστάσεις, μερικοί δεν το θέλουν. Βλέπω και στη Γερμανία τι γίνεται με τη διαδικασία της Μπολόνια και δεν είμαι τόσο αισιόδοξη ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία Αναγνώρισης συν η επαγγελματική κάρτα, συν η διαδικασία της Μπολόνια θα συνδυαστούν για να έχουμε επιτυχία. Ε, βλέπω ότι πολλά πανεπιστήμια, ε, ΑΕΗ γενικότερα, απο, ε, αποστασιοποιούνται από τη διαδικασία της Μπολόνια και θέλουν κάτι άλλο, κάτι εναλλακτικό ή το παλιό σύστημα. Άλλοι λένε όχι το νέο σύστημα είναι καλύτερο και πρέπει να το ακολουθήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι οι αντιστάσεις ήταν μεγάλες που δεν τις είχαμε φανταστεί όταν υιοθετήσαμε την οδηγία. Ο δικός σας κλάδος Ίσως ε, ε, το είδε με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και νυφαλιότητα το θέμα. Είσαστε και πρακτικοί άνθρωποι, μαθηματικά μυαλά, ε, νοημές και οι νοσοκόμοι ίσως είναι πιο θεωρητικοί ή έχουν και το στοιχείο του λειτουργήματος πιο πολύ στο επάγγελμά τους. Εγώ πάντως περίμενα περισσότερα πράγματα από την εφαρμογή του συστήματος, γιατί δεν περίμενα να είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα. Είμαστε εδώ επειδή ακριβώ υπάρχουν δυσκολίε όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα μετά την υιοθέτηση τη οδηγία και πρέπει να προχωρήσουμε. Υπάρχει σκεπτικισμό και υπάρχουν αφιβολίε, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Κυρία Πέντερσεν, λοιπόν, έχετε εδώ ένα συγκεκριμένο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσετε. Θα σα δώσω κάποια λεπτά, όπω και στον κύριο Φούξ, και επειδή έχουμε τηρήσει τον χρόνο μας. Κύριε Τίτσε, μπορεί να θέλετε κι εσείς το λόγο, γιατί στη συνέχεια έχουμε για τον κύριο Μπαρνιέ τον Επίτροπο. Να ακούσουμε και τη δική σας άποψη όσον αφορά αυτά που πάθηκα μέχρι τώρα. Η κυρία Πίτερσεν πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που άκουσα για την γραπτή δήλωση ανταποκρίνονται σε αυτά που βρήκαμε στην μελέτη. Δηλαδή, οι χώρες μέλη φαίνεται να χρησιμοποιούν την γραπτή δήλωση ως ένα είδος προτύπου τη στιγμή που η αρχική βούληση ήταν για επιλεκτική χρήση, ad hoc. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον ή χρήσιμο, ενδεχομένω και απαραίτητο όπως είπατε κι εσείς, στον τομέα των ιατρικών επαγγελμάτων και εδώ συζητήσαμε ένα παράδειγμα όπου αναφέρθηκε αυτό ως ανάγκη διαφορετικά το σύστημα ελέγχου ή εποπτείας στην συγκεκριμένη χώρα μέλος δεν μπορούσε να εφαρμοστεί εκτός και αν χρησιμοποιόταν η γραπτή δήλωση σε αυτή την περίπτωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φούξ, μήπως θα θέλατε να ολοκληρώσετε αυτό το πρώτο μέρος. ich bin der Meinung, ich... Πιστεύω, αναφερόμενο σε εσά κυρία Βάιλερ, μιλώντας για τους μηχανικούς, στη Γερμανία η διαδικασία της Μπολόνια ε, εφαρμόζεται στους μηχανικούς κατά 98%. Όχι γιατί εργάζονται σε όλο τον κόσμο και ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει ε, ένα παρόμοιο σύστημα στο 80% των χωρών για το δικό μας τον κλάδο. Ε, οπότε δεν ξέρω τόσο πολύ για τα άλλα επαγγέλματα και τις ε, ανώτατες σχολές. Εγώ είμαι πάντως πιο αισιόδοξη από εσά. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν γιατί ε, είναι σημαντικό να γίνεται μια αρχή που θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Επίσης είναι σημαντικό και εσείς στο Κοινοβούλιο να ασκήσετε την πολιτική σας ε, πειθό και ισχύ για να ακολουθήσουν όχι τόσο για τα πανεπιστήμια, όσο για τους νέους ανθρώπους που δεν θα έχουν αλλιώς ένα προσανατολισμό. Αν δεν ασκηθεί από τους πολιτικούς η απαραίτητη πίεση υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης, αυτή θα αποτύχει. Γι' αυτό λοιπόν η έκκληση μου και είναι το τελευταίο που θα πω, Σα παρακαλώ να ασκήσετε την επιρροή σα ούτω ώστε η μεταρρύθμιση τη Μπολόνια να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να μην κολλήσουμε στα μισά του δρόμου γιατί θα χάσουν τον προσανατολισμό του οι νέοι και δεν θα, κερδίσουμε τίποτα. Αντίθετα θα έχουμε καταστρέψει πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τίτζ. Θέλετε σε αυτό το σημείο της συζήτησης να λάβετε το λόγο εσεί που είχατε εργαστεί τόσο πολύ σε αυτό το κοινό μα σχέδιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θα είμαι πολύ σύντομο, επειδή θα μιλήσει αυτό το θέμα αργότερα ο Επίτροπο Μπαρνιέ. Να αναφέρω μόνο ένα σημείο γιατί η διαδικασία της Μπολόνια και η οδηγία αυτή αναφέρθηκαν επανειλημμένα. Πρόθεσή μας είναι σύντομα να ξεκινήσουμε μία μελέτη, εξωτερική μελέτη, για την διάδραση μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών διαδικασιών. Αυτό είναι το μόνο σημείο που θα ήθελα να σας κοινοποιήσω. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε στη συνέχεια από τον Επιτροπό μου. Sur euh, Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Αντώνιο Κορέα Κάμπους. Θα ήθελα η Κομισιό να λάβει το λόγο. Όμως αυτό που θα πω είναι κάτι το οποίο είναι κοινό σε όλες τις χώρες και τις αφορά. Όπως υπόθηκε εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούμε μια υποβάθμιση της διαδικασίας της Μπολόνια. Πολλά πανεπιστήμια δεν είναι ικανοποιημένα με την διαδικασία της Μπολόνια και ήδη υπάρχουν διακρίσεις όταν έχουμε αιτήσει για εργασία διακρίσεις σε πτυχία πριν Μπολόνια και μετά Μπολόνια. Αυτό σημαίνει σε αρκετές χώρες. Τα μηνύματα λοιπόν είναι πάρα πολλά που έχουμε. Και ο Σύλλογος των Μηχανικών στην ε, Πορτογαλία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα είδος μηχανισμού φιλτραρίσματος, δηλαδή να κάνει ένα τεστ, κάποιες εξετάσεις για την εγγραφή στον ε, επαγγελματικό σύλλογο, κάτι το οποίο σε τελική ανάλυση κάνει λιγότερο ευέλικτη και αποτρέπει και την ανάγκη της κινητικότητας και των γνώσεων. Βεβαίως αυτή η δικασία πάντοτε περιλαμβάνει και ένα στοιχείο επίμαχο, δηλαδή προσφυγές κλπ. Αλλά νομίζω ότι αυτό αφορά από τη φύση του περισσότερο τα ιατρικά επαγγέλματα. Και άκουσα πριν από λίγο ότι η Κομισιόν ετοιμάζει κάποιε μελέτε. Ενδεχομένω λοιπόν στι μελέτε αυτέ η Κομισιόν θα μπορούσε να κοιτάξει από διαφορετική σκοπιά το πρόβλημα. Γιατί συνήθω ε, εξετάζουμε μόνο την ασφάλεια των ασθενών ή άλλα συναφή ζητήματα, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσουν και οι φραγμοί και τα εμπόδια όσον αφορά την κινητικότητα των επαγγελματιών. Γι' αυτό ακριβώς και τα, και τα πανεπιστήμια αλλά και οι επαγγελματικές ε, ε, οργανώσεις αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουν. Να συνεχίσω να σταματήσω. Κοιτάξτε, είμαστε στο δεύτερο τμήμα, λέει η πρόεδρο, Γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να δω αν έχετε κάτι για το πρώτο τμήμα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο τμήμα, μπορείτε πάλι να λάβετε το λόγο. Κύριε Ρίσνερ, θέλετε πολύ σύντομα να πείτε κάτι. Πολύ σύντομα, συμφωνώ με τον δόκτορα Φούξε. Μια σύντομη παρατήρηση να προσθέσω. Όλη αυτή τη ρύθμιση δεν τη στηρίξουμε μόνο στη διαδικασία της Μπολόνια, γιατί τα επόμενα δέκα χρόνια θα εξακολουθούμε να έχουμε μηχανικούς που δεν θα έχουν περάσει από τη διαδικασία της Μπολόνια. Πώς σας φαίνεται αυτό. Α, πολύ ωραία. Σύντομη απάντηση. Ναι, εμείς τις λάβαμε υπόψη αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό χρειάζονται οι εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή ε, των Ειδικών που γνωρίζουν και τα παλιά συστήματα και την Πολόνια. Οπότε βεβαίως λαμβάνεται υπόψη αυτό. Ωραία, θα ξεκινήσουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας και θα ασχοληθούμε περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη και ε, τα όσα είπαν και οι παρεμβαίνοντες ε, στους ε, εκπροσώπους του τομέα της υγείας. Θα δώσω σε λίγο το λόγο στον κύριο Φουρτουή, ο οποίος, ο οποίος εκπροσωπεί ε, την, ε, ε, τους φαρμακοποιούς της Γαλλίας. Ε, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα των αναγνωρίσεων των προσόντων και μετά θα δώσω το λόγο στον ε, καθηγητή Τόνι Χέιζελ ο οποίος είναι πρόεδρος ε, της οργάνωσης νοσηλευτριών, νοσηλευτών, νοσηλευτριών και μεών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο καθηγητής ε, ε, Χέιζελ επίσης, ε, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής, έχει αναλάβει εξ ονόματος της Επιτροπής να συλλέξει τα εθνικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φορτουή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρεμβαίνω σε ένα σημείο της συζήτησης όπου ήδη έχουν αναφερθεί τα προβλήματα του ε, τομέα ε, υγείας ε, και επομένως μπορεί να πω κάποια γενικά θέματα τα οποία μετά να συζητηθούν ενδελεχώς. Πρώτα θα σας μιλήσω για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα αναφερθώ στις ε, ε, εισηγήσεις που αφορούν εμπειρίες φαρμακοποιών, αποτελέσματα μελετών ε, τα οποία, και τα αποτελέσματα των μελετών τα οποία έχουμε διεξάγει κυρίως στη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου γιατί δουλέψαμε τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο για το θέμα αυτό. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο, βεβαίω, το υπενθυμίσατε κι εσείς, εμείς βρισκόμαστε στα πλαίσια της ε, οδηγίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσώπων 2005-36 ε, σε, ε, η οποία υπενθυμίζω ότι περιλαμβάνει τι 15 υφιστάμενε οδηγίες, 5, κατηγορίε κατηγορίες υγείας, γιατρούς, χειρουργούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, και μέσα. Πρέπει να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι στα πέντε χρόνια θα υπάρξει αναθεώρηση, πιθανή αναθεώρηση και με πάση περιπτώσει επανεξέταση της οδηγίας και των μέχρι τότε ε, αποτελεσμάτων. Ε, βεβαίως εμείς ε, ε, θέλουμε να μεταφέρουμε την αξιολόγηση ε, και ευχαριστώ όσους αναφέρονται στο θέμα αυτό και όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό και αυτή η πρώτη αξιολόγηση που έχει γίνει σε μερικές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να δούμε εάν υπάρχει μια συνολική ευρωπαϊκή δομή η οποία θα συγκεντρώνει τις αρμόδιες αρχές των διαφόρων επαγγελμάτων και αν μπορεί να γίνει και μια αξιολόγηση ένα επάγγελμα. Γιατί βεβαίως εγώ θα αναφερθώ σήμερα στους φαρμακοποιούς. Ποιες ε, είναι ε, οι ε, εισηγήσεις, ποιες είναι οι εκθέσεις σε βάση των εμπειριών μας. Ε, έλαβαν χώρα τρεις ε, συνεδριάσεις, οι οποίες οργανώθηκαν στις 7 Ιουνίου η πρώτη και μέχρι το Σεπτέμβριο η τελευταία. Εργαστήκαμε βάσει ενός προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο βασιστήκαμε έτσι ώστε να εκπονήσουμε ερωτηματολόγιο. Ξαναβρεθήκαμε λοιπόν στις 9 Ιουλίου πάντα του 2010 έτσι ώστε να συζητήσουμε τα κυριότερα θέματα, τα θέματα κλειδιά, τα οποία μας φαίνονται πιο σημαντικά, δηλαδή η εγκατάσταση, ε, η προσωρινή παροχή υπηρεσίας, ε, η κατάρτιση, αλλά και η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες αρμόδιες αρχές. Συναντηθήκαμε και μια τρίτη φορά όμως για να δούμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι μεγάλες τάσεις ε, που διαφαίνονται οι προτάσεις ε, αυτές έγιναν από τις αρμόδιες αρχές. Ε, εμείς επίσης ε, ήρθαμε σε επαφή με τις 27 αρμόδιες αρχές για τους φαρμακοποιούς και πρέπει να σας πω ότι αυτές οι 18 ε, εκθέσεις ε, για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κυριότερα αποτελέσματα είναι βεβαίως θα πρέπει να αναφερθούν σε μια πρώτη φάση. Ε, το πρώτο που θέλουμε είναι να διευκολύνουμε την κινητικότητα των επαγγελματιών της υγείας και βεβαίω μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο ε, παρακαλώ πολύ το λέω στον υπεύθυνο των, ε, ε, των slides ε, δεν θέλω να πω βεβαίως πάρα πολλά, ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω έτσι ώστε να αφήσω και χρόνο ε, τους, στις ερωτήσεις. Έλεγα όμως ότι τα κυριότερα αποτελέσματα είναι ότι βλέπουμε ότι πρέπει να βελτιωθούν και να διευκολυνθούν οι συνθήκες της κινητικότητα των επαγγελματιών της ε, υγείας. Ακούσαμε ε, ορισμένα προβλήματα που έχουν υπάρξει λόγω της κινητικότητας στην ε, Μεγάλη Βρετανία και επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει καλή αναγνώριση. Βεβαίως τα επαγγελματικά λάθη υπάρχουν πάντα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι υποπίπτουν σε λάθη κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ε, στην χώρα τους ε, και που ε, τους απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πάνε σε μια άλλη χώρα και να ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση, νομίζω ότι εδώ το πράγμα είναι αρκετά απλά η αυτόματη αναγνώριση φαίνεται ότι είναι επιτυχής και για τις αρχές και για τους ε, φαρμακοποιούς. Τα θέματα λοιπόν διευθετώνται με τον τρόπο αυτό. Ε, ξέρετε μερικές φορές έχουμε τη τάση να μιλάμε μόνο για αυτά που δεν πάνε καλά. Όταν κάτι πάει καλά τότε δεν έχουμε πρόβλημα ε, και δεν το ε, συζητάμε. Σε γενικές γραμμές λοιπόν εδώ πάνε όλα καλά Και νομίζω λοιπόν ότι για την περίπτωση ε, για την περίπτωση των φαρμακοποιών τα πράγματα είναι καλά. Ε, νομίζω ότι ε, για την ώρα έχουμε ένα καλό σύστημα αναγνώρισης το οποίο είναι σχετικά καινούργιο, δεν υπήρχε πριν. Έχουμε μάλλον περιορισμένο αριθμό προβλημάτων, αλλά βεβαίω η εμπειρία μα δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Φαίνεται ότι ο τρόπο πάντω λειτουργία είναι αρκετά ικανοποιητικό. Το θέμα της το θέμα της ε, κατάρτισης, ε, της διάρκειας κατάρτισης μας προβληματίζει λίγο περισσότερο. Ε, το περιεχόμενο της κατάρτισης, σύμφωνα με τις απαντήσεις που είχαμε από τις αρμόδιες αρχές, είναι μάλλον ικανοποιητικό. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να υπάρξει εναρμόνιση όσον αφορά τις, τα στάζ, όσον αφορά δηλαδή τις, τα προγράμματα, τα προγράμματα κατάρτισης ε, μας ενδιαφέρει στη διάρκεια αυτού του στάζ να ε, μαθαίνει ο φαρμακοποιός τις τεχνικές ε, του επαγγέλματος. Ε, επίσης, θα πρέπει να, να δούμε όχι μόνο πόσο κρατάει η κατάρτιση αλλά πόσα μαθήματα, πόσες ώρες μαθημάτων προβλέπονται πραγματικά και βεβαίως εκεί εισέρχεται και το πρόβλημα της γνώσης της γλώσσας ε, της ε, χώρας ε, υποδοχής. Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης του περιεχομένου κατάρτισης των φαρμακοποιών ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη και όσον αφορά την κοινωνία και όσον αφορά ε, τα νέα επαγγελματικά προσόντα ε, και στην θεραπευτική κοινότητα. Στην Γαλλία, ας πούμε, το ΕΣΠΕΑΖΕ άλλαξε τις προϋποθέσεις και τις αρμοδιότητες των φαρμακοποιών. Υπάρχει, υπάρχουν εξελίξεις και όσον αφορά τα νομικά κείμενα και όσον αφορά τις διάφορες χώρες και επομένως θα πρέπει η κατάρτιση που θα δίδεται στο προσωπικό προσωπικού να είναι αντίστοιχη ε, με τις ε, ε, όποιες εξελίξεις υπάρχουν στον τομέα της υγείας γενικότερα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι η διαβίου κατάρτιση. κοιτάξτε, εγώ πήρα το πτυχίο μου το 1970. Εάν από τότε δεν είχα λάβει οποιαδήποτε κατάρτιση, οποιαδήποτε περαιτέρω εκπαίδευση καταλαβαίνετε ότι ε, θα είχα μείνει πάρα πολύ πίσω στο επαγγελμά του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα ε, με εκπαίδευσης όχι μονάχα στην χώρα του φαρμακοποιού ή στη χώρα άσκησης ε, του επαγγελματο του φαρμακοποιού αλλά και σε άλλες χώρες εάν θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα κατάρτιση το οποίο είναι καλό και είναι σε μια άλλη χώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε, να βοηθήσουμε την κινητικότητα. Τώρα, ε, δύο-τρία σημεία ήθελα να πω ακόμα. Όσον αφορά την συνεργασία λοιπόν ε, μεταξύ των ε, αρμοδίων αρχών, είπαμε ότι οπωσδήποτε οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Είπαμε και προηγουμένως ότι σε γενικές ε, γραμμές ε, ε, διαπιστώνουμε ικανοποίηση των αρμοδίων αρχών όταν χρησιμοποιούν το, το πρόγραμμα των της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την, το πόρταλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επίσης λυπούμεθα γιατί όλες οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμα ε, υποβάλει τα προγράμματά τους. Επομένως μπορούν να γίνουν ακόμα περαιτέρω ε, βελτιώσεις και μάλιστα με τρόπο εργονομικό. Για να ολοκληρώσω λέω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίσουμε την αξία Τη της συνεργασίας, την αξία της κινητικότητας. Ε, πρέπει να πω ότι από κάποιες χώρες είχαμε πάρα πολύ ικανοποιητικέ απαντήσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα. Ε, αυτή η Ευρωπαϊκή Κάρτα πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιώσει και τη συνεργασία και το συντονισμό και να δώσει προστιθέμενη αξία στην αναγνώριση των διπλωμάτων, αλλά βεβαίως απαραίτητο είναι να ορίσουμε καλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δίδεται αυτή η κάρτα. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρέπει οπωσδήποτε να σκύψει περισσότερο πάνω από αυτό το πρόγραμμα στα πλαίσια της αναθεώρησης της ε, οδηγίας που αναφέραμε και στην αρχή. Αναφερθήκαμε προηγουμένως ας πούμε στην διαβίου κατάρτιση. Πιστεύουμε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Κάρτα θα μπορούσε να βοηθήσει ιδιαιτέρως, να διευκολύνει ιδιαιτέρως ε, αυτήν την διαβίου κατάρτιση. Επίσης ε, να δίνει ε, πρόσβαση στα, στους ιατρικούς φακέλους Αυτά ήθελα να σας πω. Βεβαίως ακόμα συνεχίζουμε. Είναι πολύ λίγος ο καιρός ε, κατά τον οποίο ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανάλυση μας. Βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε την συνεργασία μας με τις αρμόδιες αρχές ε, να πω εν συμπεράσμα ότι θεωρούμε ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καινοτόμα. Ε, να πούμε επίσης ότι ε, όσον αφορά τους ε, φαρμακοποιούς εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε επί της ουσίας ε, το κουρίκουλουμ, τα μαθήματα και την κατάρτιση την αρχική των φαρμακοποιών θα πρέπει να ξαναδούμε την διαρκή κατάρτιση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων αρχών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται αυτές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης εργαλεία όπως αυτή η Ευρωπαϊκή, Τράπεζα, ε, ε, ε, Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό εάν ακολουθήσουμε το πνεύμα μέσα στο οποίο αυτή δημιουργήθηκε. Αυτές είναι λοιπόν οι κεντρικές γραμμές, οι κεντρικοί άξονες στους οποίους έχουμε καταλήξει ε, όσον αφορά την μελέτη του θέματος από πλευράς των φαρμακοποιών. Ε, πρέπει να σας πω ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και λίγο καιρό. Αρμόδιες αρχές, εκπρόσωποι των φαρμακοποιών, εκπρόσωποι επαγγελματιών κλπ. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την εξαιρετικά επικοδομητική εμπειρία την οποία, ε, μας, ε, ε, την οποία μοιραστήκατε μαζί μας και έχει δίκιο η Μπάρμπαρα όταν λέει ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε ενθουσιώδεις, πρέπει να με μεγάλο κέφι και μεράκι να ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χέιζελ, ο οποίος εκπροσωπεί τις νοσηλεύθερες και τις ΜΕΣ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτή την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα, το οποίο θεωρώ μια τιμή. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Όπω γνωρίζετε όλοι, αυτή η διαδικασία αποτελεί το, την πρώτη φάση διαβούλευση τη ανθεώρησης τη οδηγία και αποσκοπεί στο να παράσει πληροφορίε στην Κομισιόν όσον αφορά την εφαρμογή τη οδηγία σε διάφορε χώρε μέλη. Το NMC με χαρά αποδέχτηκε την εργασία συντονισμού όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών για τις νοσοκομές και τις ΜΕΕΣ. Αποτελούμε ένα ανεξάρτητο ρυθμιστικό σώμα και είμαστε το μεγαλύτερο ρυθμιστικό σώμα στον κόσμο με πάνω από 650.000 άτομα στο μητρό μας. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με το αντίστοιχο σώμα το γαλλικό που συντόνισαν τις ε, απαντήσεις όσον αφορά τις ΜΕΕΣ. Η διαδικασία διαβούλευσης ακολούθησε ένα κοινό ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από κοινού με την Κομισιόν και τροποποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Όπως είδατε κάθε δίκτυο είχε τρεις συναντήσεις και χαρήκαμε με τις θετικέ ανταποκρίσεις που είχαμε για συμμετοχή και αυτό ιδιαίτερα μετά από πολύ σύντομη ειδοποίηση ή χωρίς πολύ χρόνο για ειδοποίηση. Ως αποτέλεσμα είχαμε 26 εκθέσεις για τις, για τις νοσοκόμες και 24 για τις ΜΕΣ. Και νομίζω ότι οι περισσότερες από αυτές τις εκθέσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές. Όπως ε, θα περιμένατε υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις στον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας και σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται στον, ε, στην ποικίλουσα φύση των αρμοδίων αρχών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία ανέκυψαν κοινά για όλη την Ένωση και τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Η γραφική έκθεση του NMC είναι ήδη διαθέσιμη για αυτά τα θέματα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Το πρώτο θέμα που εντοπίσαμε ήταν το θέμα της ελάχιστης κατάρτισης η εκπαίδευση και πάλι θα γνωρίζετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με πριν από τρει ε, δεκαετίε και τώρα όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι ΜΕΣ και οι νοσοκόμε έχουν νέου ρόλου και νέε ευθύνε. Όλο και περισσότερο οι νοσοκόμε και άλλα ιατρικά επαγγελμάτα καλούνται να παρανεύουν βάσει κάποιων ενδείξεων και δεν θα πρέπει θα πρέπει να αναπτύξουμε νέες μεθόδους εκμάθησης που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις εξελίξεις. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή οι ΜΕΕΣ και οι νοσοκόμες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις ανταποκρινόμενες με τον μέγιστο δυνατό ή καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις αυτές. Το θέμα της ανταλλαγή πληροφοριών. Είχαμε διάφορες προσεγγίσεις οι οποίες ε, είχαν και αντίκτυπο όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων στις χώρες μέλη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε συμφωνία και το ακούσαμε και από άλλους ότι ο μηχανισμός IMI θα πρέπει να επεκταθεί στα τομεακά ε, επαγγέλματα, ιδιαίτερα τα επαγγέλματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών. Τέλος, το θέμα της λογιστικής επάρκειας. Από τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις διάφορες αρμόδιες αρχές είδαμε ότι αυτό αποτελεί κυρίως ευθύνη και αρμοδιότητα του εργοδότη. Παρ' όλα αυτά, από τις 26, 13 εκθέσεις περιλάμβαναν σαφείς ενδείξεις όσον αφορά τις, ε, τα γλωσσικά προσόντα νοσοκόμων και μεών οι οποίες ε, πηγαίνουν να εργαστούν σε χώρα εκτός της δικής τους. Ελπίζω ότι αυτή η πολύ σύντομη παρουσίαση των κοινών σημείων να σας βοηθήσει ώστε να γίνει σωστά αυτή η πενταετής αναθεώρηση της οδηγίας και να επιθυμίσω και πάλι στα μέλη ότι η γραπτή μας μελέτη με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Ευχαρίστως θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Euh, Ευχαριστώ. Διαπιστώνω ότι είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο. Καλό τους βουλευτές από άλλες χώρες και που ήρθαν να ακούσουν να τοποθετηθούν, να λάβουν το λόγο γιατί είναι σημαντικό να ακούσουμε την απόψή τους. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σπύρο Ταλιαδούρο ο οποίος έρχεται από την Ελλάδα και ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ε, και να παρακαλέσω τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τις λάβουν υπόψη τους. Ε, είναι σαφές ότι στόχος της οδηγίας είναι η διευκόλυνση της ενδοκινοτικής κινητικότητας των εργαζομένων και της παροχής υπηρεσιών. Υιοθετήθηκε για την εξάλληψη των εμποδίων της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των υπηρεσιών. Αφορά πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Όμως, μετά την εφαρμογή στην Ελλάδα από το Μάιο της οδηγίας, στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 90% αυτών που κάνουν χρήση αφορά Έλληνες φοιτητές εξωτερικού οι οποίοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις αυτές για να αποφύγουν τον εθνικό φορέα ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων ξένων πανεπιστημίων. Συμφωνούμε απολύτως ότι θα πρέπει να υπάρχουν εργαλεία που θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά τα εργαλεία αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο που να ακυρώνουν ρυθμίσεις που αφορούν τους πολίτες των κρατών μελών. Πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες. Δεύτερον, η αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχει επιτευχθεί σε ορισμένα επαγγέλματα του ιατρικού χώρου και των αρχιτεκτόνων δεν θα πρέπει αυτόματα να επεκταθούν και σε άλλα επαγγέλματα. Γιατί ανάμεσα στα κράτη-μέλη υπάρχει συχνά τεράστια απόκληση μεταξύ των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και είναι δύσκολο πολλές φορές να υπάρξει αυτόματη αντιστοίχηση. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή που στην Ελλάδα για την άσκησή του απαιτείται πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ σε άλλα κράτη-μέλη αρκεί ή να είναι κάποιος απόφυτος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τρίτον, η απλή γνωστοποίηση μόνο των επαγγελματικών στοιχείων του παρέχοντος υπηρεσία χωρίς αξιολόγηση και έλεγχο των γνώσεών του δεν διασφαλίζει το εάν οι γνώσεις αυτού που κάνει την αίτηση είναι επαρκής και αντιστοιχούν στα εθνικά δεδομένα. Τέταρτον, ελέγχθηκε πριν, θεωρώ ότι απαιτείται να υπάρχει καλή γνώση της γλώσσας υποδοχής και να υπάρχει έλεγχος κατά την εξέταση του φακέλου. Τέλος, η τροποποίηση, η συνολική τροποποίηση της οδηγίας ίσως σήμερα να είναι ακόμα πρόωρη. Ίσως θα πρέπει να προηγηθεί κάποια εμπειρία ακόμα, να έχουμε κάποια αξιολόγηση της εφαρμογής του. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη μελέτη. Και αυτό το λέω γιατί στην προσπάθειά μας να γίνουμε μια πραγματική ένωση χωρίς σύνορα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, θα δώσουμε τον ε, λόγο στον κύριο Φιλίππο Μπουρίκο από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι στην αναθεώρηση της ε, οδηγίας ε, ότι η αναθεώρηση πάνω της οδηγίας μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για να ε, δούμε, να δώσουμε νέες απαντήσεις στα προβλήματα τα οποία προέκυψαν και τα είδαμε ότι προέκυψαν στην, ε, στον χρόνο, στον πρώτο χρόνο εφαρμογής της οδηγίας. Δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουμε εσωτερική αγορά, κυρίως δε στην δύσκολη φάση την οποία διανύουμε με τρόπο διαφορετικό. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε βεβαίως τις τις εχθρότητες, ε, τις, τους φόβους, ε, τα εθνικιστικά κλεισίματα έτσι όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση Μόντι. Επομένως, για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφείς κανόνες. Να απαγορεύσουμε υπεκφυγές ε, ή μεθόδους υπεκφυγής από διάφορες χώρες, να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε πρότυπα ε, για όλα τα επαγγέλματα τα οποία έρχονται σε επαφή ε, με το καταναλωτικό κοινό, να ε, καθορίσουμε επίσης ελάχιστα κοινά πρότυπα για την διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από, τους, ε, από τον εκπρόσωπο των Ιταλών μηχανικών και πιστεύω ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά καλή ε, συνεισφορά ε, στην δημιουργία ενός γόνιμου κλίματος για την εφαρμογή αυτού του ευρωπαϊκού επαγγελματικού ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας που μπορεί να είναι ένας επιτεύξιμος στόχος ε, πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε εργαλεία και μεθόδους αμοιβαία αναγνώρισης επαγγελματικών προσώπων που να είναι πραγματικά πλήρης αναγνώριση. Πολύ ενδιαφέρουσες μου φάνηκαν και οι παρατηρήσεις της κυρίας Ράνμπολ ε, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα ε, στα οποία κατέληξαν εκπρόσωποι των επαγγελμάτων θεμάτων υγείας ε, κυρίως δε αυτά που ακούσαμε από τους φαρμακοποιούς, εκπροσώπους δηλαδή των φαρμακοποιών, των νοσηλευτών και των μεών με τη διαδικασία της ε, Μπολόνιας. Αυτή η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει. Αλλά και οι επαγγελματικές εμπειρίες των επαγγελματικών οργανισμών θα πρέπει να προχωρήσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Γιατί η εκπαίδευση και η επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει να συγκλίνουν μέσα από μια προσπάθεια καθορισμού ενός ευρωπαϊκού κοινού χώρου των αρμοδιοτήτων και των προσόντων και των επαγγελματικών ικανοτήτων. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύτιμη για την σκέψη που και τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι Εθνικές Κυβερνήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν και θα είναι η μεγάλη συμβολή του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να την βοηθήσει στην βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών δομών αναγνώρισης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ιδιαίτερα η τελευταία σας φράση που είναι ουσιώδης αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφά μου, στον κύριο Ζιβάν, ευρωβουλευτή, που όμως έχει ένα επάγγελμα που σχετίζεται άμεσα με τη συζήτηση αυτή. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι γιατρός όπως και άλλοι εδώ και γνωρίζω το θέμα πριν γίνω ευρωβουλευτής. Πολλά υπόθηκαν και νομίζω ότι η κυρία Βέιλερ συνόψε το θέμα προηγουμένως λέγοντας ότι Όλοι μας είμαστε πεπισμένοι ότι η εκπαίδευση στις χώρες μας αναπάγγελμα είναι καλύτερη. Και αυτό θεωρούν και οι περισσότεροι πολίτες. Και εδώ ακριβώς είναι δυσκολία, γιατί σε ένα ιδανικό κόσμο, αν το επάγγελμα ήταν ταυτόσιμο από τη μια χώρα στην άλλη, το οποίο δεν συμβαίνει όμως σήμερα, μια Βρετανίδα ε, νοσοκόμο, δεν κάνει την ίδια δουλειά καθημερινά με μια Γαλλίδα νοσοκόμο. Αν όλα τα επαγγέλματα ανταποκρινόταν στην ε, ουσία στο ίδιο λειτουργήμα και αν η κατάρτιση, η αρχική κατάρτιση ήταν ταυτόσιμη, δεν θα είχαμε λόγο να βρεθούμε εδώ σήμερα να συζητήσουμε, γιατί αλλιώ δεν θα υπήρχε ο φόβος αναγνώρισης σε μια χώρα Α της κατάρτισης εκπαίδευσης που δόθηκε σε μια χώρα Β. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή ακριβώ μα ενδιαφέρει αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ, σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθούμε εδώ σε πέντε ή σε δέκα χρόνια να ξαναδούμε το γιατί δεν λειτουργήσε η αναθεωρημένη οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε άμεσα με το θέμα της πρώτης, της ε, πρωτογενούς κατάρτισης. Δεύτερον, το πραγματικό πρόβλημα, το είπατε όλοι σας, είναι αυτός ο φόβος, ο φόβος και η αμφιβολία και η εθνική υποχώρηση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είτε ο κάθε επαγγελματίας, ο καθένας στον τομέα του θα μας βοηθήσει ώστε να βρούμε κοινά σημεία και τα, στοιχεία, και τα στοιχεία αυτά που θα μας επιτρέψουν ένας Γάλλος ιατρός να είναι εξίσου κατερτισμένος όπως ένας Ιταλός και ένας Ρουμάνος ή τότε θα έπρεπε οι επαγγελματίε να μας ε, βοηθήσουν και να τα κάνουμε αυτά ή δεν θα μας βοηθήσουν οπότε οι εθνικοί νομοθέτες θα έπρεπε να επιταχύνουν τα πράγματα μέσω μικρών εργαλείων που θα πρέπει να εφαρμόσουν εργαλεία τα οποία θα έχουν ως στόχο να καταπολεμήσουν τους εθνικούς φόβους οι εθνικοί φόβοι σε τι συνίστανται δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε συζητώντας με τους άλλους. Αν όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν τουλάχιστον εν μέρη με ταυτόσιμο τρόπο. Αν λοιπόν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτή την ταυτόσιμη εκπαίδευση, αν κάποια στιγμή πάνε στο εξωτερικό να δουλέψουν κινητικότητα καθηγητών, φοιτητών κτλ., τότε εκεί πραγματικά αυτό θα ήταν μια εύκολη τεχνική να βρούμε κάποια λύση και να αποδεχθούμε τον άλλον. Η πιστοποίηση των καθηγητών και των κέντρων εκπαίδευση είναι ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω, Πρόεδρε, μετά από αυτά που είπαν και οι μεν και οι δε, νομίζω ότι το στίχημα κυρίω είναι βεβαίω τεχνικά, αλλά κυρίω είναι ψυχολογικό. Να μην φοβόμαστε δηλαδή τον άλλον και την εκπαίδευση που κάνει στου ε, φοιτητέ του και του μαθητέ του. Παρά δηλαδή τι διαφορέ στην εκπαίδευση, από χώρα σε χώρα. Είμαι βέβαιος και πεπισμένο ότι στην Ευρώπη εξίσου όλοι λαμβάνουμε την ίδια την ίδια περίθαλψη, τη στιγμή που οι γιατροί δεν έχουν την ίδια κατάρτιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στη Βουλή των Λόρδων, η Βαρόνη Οκασίν, που είναι παρούσα εδώ και εκπροσωπεί την ε, Επιτροπή εσωτερική Αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ω Πρόεδρος της Υποεπιτροπή για την Εσωτερική Αγορά υποστηρίζουμε την ιδέα της κινητικότητα των επαγγελματιών ελεύθερη κινητικότητας σε όλη την εσωτερική αγορά. Όμως η εμπειρία στον Βασίλειο μας δείχνει το τωρινό σύστημα και η εφαρμογή του δεν είναι τέλεια, όπως ήδη ακούσαμε. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα είναι απλό, ευκολονόητο και από το κοινό αλλά και τους επαγγελματίε, θα είναι διαφανές, θα είναι αξιόπιστο, δεν θα είναι ακριβό και δεν θα είναι εύκολο να έχουμε απάτες και εξαπάτες σε αυτό το σύστημα όπως ακούσαμε προηγουμένως ε, τα ιταλικά παραδείγματα. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να είναι δυνατότητα στις χώρες μέλη να διασφαλίσουν στους πολίτες άλλων χωρών τη δυνατότητα ελεύθερης εργασίας. Αυτό είναι απαραίτητο. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει να περιλάβουμε και το θέμα της γλώσσας και της γλωσσικής επάρκειας. Θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές σε κάθε χώρα μέλος να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους ώστε όπως έδωσε το παράδειγμα κυρία Στήλε από το Ηνωμένο Βασίλειο οι ισπανικές αρχές να κοινοποιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο περιπτώσει όταν κάποιος γράφεται ας πούμε από το ιατρικό μητρό θα πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς ακριβώς οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να συνεργαστούν και νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία το γεγονό ότι θα πρέπει να κινηθούν και να εργαστούν ελεύθερα οι επαγγελματίε, ακολουθώντα όλε αυτέ τι διαδικασίε με τι απαραίτητε δικλείδε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο λόγο τώρα στον κύριο Μιχαήλ Παντούλα, ο οποίο είναι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκτός μικροφώνου. Μικρόφωνο ανοίξτε. Κύριε Πρόεδρε, μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία και αφού χρειάστηκε να ξεπεράσουμε πολλά προβλήματα, η Ελλάδα, όπως ακούσατε και από τον κύριο Ταλιαδούρο, το Μάιο του 2010 με ρυθμιστική πράξη, δηλαδή με έκδοση προεδρικού διατάγματος, αποφάσισε την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ήταν μία από τις προτεραιότητες της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία, όπως γνωρίζετε πολύ εδώ μέσα στην αίθουσα, διετέλεσε και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή, όπως έχω δει, ίσως να κάνω λάθος κυρία Πρόεδρε, δεν έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα της εσωτερικής αγοράς του Ιουλίου του 2010. Το γεγονός αυτό δεν απεικονίζει την πραγματική εικόνα στην πρόοδο της χώρας μου στο συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς και δεν υπονοώ καμία σκοπιμότητα, ίσα ίσα τιμώ το έργο της Επιτροπής και εσάς προσωπικά. Το επισημαίνω απλώς για να συμπεριληφθεί στον επόμενο πίνακα. Είναι ε, αυτονόητο ότι δεν θέλω να δικαιολογήσω την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση όμως της Ελλάδας κινείται με σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να υπερβούμε τα προβλήματα. Σήμερα κινούμαστε σε τροχιά εφαρμογής σε όλα τα πεδία με βάση τις εξαντλητικά λεπτομερείς διατάξεις του προεδρικού διατάγματος που προανέφερα, ώστε να υπερβούμε τη διοικητική, συντεχνιακή ή άλλου είδους γραφειοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς ότι δεν υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Μέρος αυτών των προβλημάτων τα εξέθεσε με ενάργεια η κυρία Μπόλντι από την Ιταλία. Είναι επισημάνσεις που κατέθετε πάντοτε η Ελλάδα. Εμείς και η Ιταλία είμαστε σε μια περιοχή που αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα που ενδεχομένως να είναι άγνωστα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ό,τι ανέφερε η κυρία Μπόλντι θα ήθελα να προσθέσω έναν προβληματισμό σε σχέση με τους μηχανικούς. Υπάρχουν πολυτεχνία σε ευρωπαϊκές χώρες όπου στο πρόγραμμα σπουδών τους δεν συμπεριλαμβάνεται μαθήματα για παράδειγμα αντισυσμικής προστασίας των κτηρίων επειδή αυτές οι χώρες δεν βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο. Πώς λοιπόν θα ελεγχθούν οι γνώσεις των ενδιαφερομένων σε αυτό το επίπεδο που είναι κρίσιμο σημείο για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Στην ε, ενσωμάτωση της οδηγίας η Ελλάδα θεώρησε ότι τα ε, ε, επαγγέλματα του αρχιτέκτονα, των γιατρών, των μεών, των νοσοκόμων, των φαρμακοποιών αναγνωρίζονται αυτόματα, χωρίς καμία διαδικασία. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα εκεί. Αναφέρθηκε ήδη από διάφορους ομιλητές το πρόβλημα της γνώσης της γλώσσας των χωρών υποδοχής και δεν θέλω να το επαναλάβω. Κλείνοντας κυρία Πρόεδρε, θέλω να τονίσω τη διάθεσή μας να συμβάλλουμε με θετικό και γόνιμο τρόπο στην όλη διαδικασία από εδώ και πέρα η εμπειρία της εφαρμογής είναι βέβαιο ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ο διάλογος και με τα εθνικά κοινοβούλια αξίζει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος να προχωρήσουμε σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε διάλογο και στο μέλλον μεταξύ... Ε, <laughs> εδώ μάλλον ε, θα έχετε πάλι ελληνικά θα ακούσετε από τον κύριο Τριανταφυλλίδη όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο σημεία να θίξω. Το πρώτο αφορά την απασχόληση και τα εργασιακά δικαιώματα και δεδομένου ότι η διακίνηση των εργαζομένων διασυνοριακά είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης, και ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι κύριο συστατικό αυτής της πολιτικής, ερωτώ πώς η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων συνδέεται με τα διάφορα καθεστώτα συλλογικών συμβάσεων που ισχύουν στα 27 κράτη-μέλη. Γιατί φοβούμε ότι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων θα έχει επιπτώσει στα εργασιακά δικαιώματα και θα πρέπει να βρούμε ρύθμιση ώστε να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εργασιακό περιβάλλον κατά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τις λανθασμένες διασυνοριακές πρακτικές ή παρανομίες. Ε, στις μεθόδους προστασίας από αυτές τις λανθασμένες πρακτικές ποιο νομικό καθεστώς θα δεσμεύει τον επαγγελματία που παρανομεί διασυνοριακά Αφενός υπάρχει ρύθμιση που να αποτρέπει όσους έχουν στο βιογραφικό τους παρανομίες και αμέλειες σε ένα κράτος μέλος να εργαστούν σε άλλο. Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις διασυνοριακών παρανομιών, υπάρχει ευρωπαϊκή ομπρέλα που να καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις ή διέπεται εθνικά και πώς διασφαλίζεται η ορθή νομική διαδικασία. Πριν δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες ε, που θα απαντήσουν σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που θέσατε, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γιαζίνσκι, ο οποίος ε, έρχεται από την Πολωνία, εκπροσωπεί την Βουλή της Πολωνίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Pani Przewodnicząca. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Είμαι Πολωνός και προκειμένου περί της εφαρμογής της οδηγίας στην Πολωνία ε, δεν ε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εγώ κάτι άλλο θέλω να αναφέρω. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές στα προσόντα ε, παίζουν ρόλο οι διαφορετικές ε, παραδόσεις. Αυτό ισχύει και για τους μηχανολόγους μηχανικούς, όπως είπαμε. Αλλά βέβαια η εργασία ενός μηχανικού μπορεί να μην επηρεάζει τόσο πολύ την υγεία και τη ζωή ενός ανθρώπου. Ενώ ε, τα ιατρικά επαγγέλματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει εξομοίωση, αλλά δεν μπορούν να καταργηθούν κάποιες διαφορές μεταξύ επαγγελμάτων. Καλό είναι που εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι τα αποτελέσματά μας όλο και βελτιώνονται. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, ομιλητές μας αν οι κυβερνήσεις και οι επαγγελματικές οργανώσεις ακολούθησαν διαφορετική προσέγγιση κατά την απάντηση κάποιων ε, ερωτημάτων. Μπορεί η κυβέρνηση τα ιατρικά θέματα να τα προσεγγίζει διαφορετικά αφού αφορούν την ζωή και την υγεία των ανθρώπων και οι επαγγελματικές οργανώσεις μπορεί πάλι να έχουν διαφορετική θεώρηση του προβλήματος. Μπορεί οι τελευταίες να θεωρούν ότι είναι το πιο σημαντικό να περιοριστεί ο ανταγωνισμός. Στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα είναι και αυτό σημαντικό. Ε, για από τους ε, μηχανικούς ε, εξαρτάται πόσο θα προχωρήσει η οικονομία ε, και πώς θα εναρμονιστούν οι κανόνες σε αυτό το τομέα στην Ευρώπη ενώ στους γιατρούς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να δώσουμε απαντήσεις θα πάρουν το λόγο οι εμπειρογνώμονες γιατί νομίζω μόνο δύο ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Στίτλερ και μετά τον κύριο Κορέα Κάμπος. Και μετά οι εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά τον προαλήσαντα σκεφτόμουν κατά πόσο η η βιομηχανία η κατασκευαστική είναι πιο επικίνδυνη όσον αφορά την υγεία αν σκοτωθεί ένας εργαζόμενος υπάρχουν διαφορές βέβαια όσον αφορά την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τα προσόντα αλλά νόμιζα ότι μέχρι τώρα υπήρχε πλήρης διαφορά μεταξύ του τομέα της υγείας και άλλων τομέων όμως εδώ θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά και ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το γεγονός ότι τα προσόντα και η κατάρτιση των ε, μηχανικών είναι και μέσω ίντερνετ. Το ίδιο και με τους φαρμακοποιούς. Τι γίνεται με το ενδεχόμενο μιας ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας και το ενδεχόμενο ανταλλαγής αυτής της κάρτας ηλεκτρονικά. Υπάρχουν διαφορές για τους διάφορους επαγγελματικού τομείς, νοσοκόμες κτλ. Ακούσαμε για τις βαλτιστές πρακτικές και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό βέβαια το θέμα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Όμως έχουμε και το θέμα των προδιαγραφών σε σχέση με το τι κάνουν οι νοσοκόμες στη Γαλλία ή στην Αγγλία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημείο συζήτηση αν θέλετε. Θα μπορούσε να γίνει και έχει σχέση με τη συζήτηση για την τυποποίηση. Και βεβαίως αφορά και το θέμα αυτό της επαγγελματική ηλεκτρικής κάρτας που θα μπορούσε κανείς να θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κορέα Κάμπος. Ευχαριστώ, Μπερναντέτ. Η χώρα μου έχει γύρω στο 15 100 ξένων γιατρών και νοσοκόμων. Οπότε όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη μιλάμε για παρουσία επαγγελματιών αρκετά σημαντική. Για το μέλλον ίσως να χρειάζεται να έρθουν περισσότεροι αλλά υπάρχουν φραγμοί στην μετακίνησή τους. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι αυτοί ξεκινούν με διαφορετικές προϋποθέσεις ή διαφορετικές, ε, διαφορετικούς στόχους, αλλά αντιμετωπίζουν διαφορετική κατάσταση όταν φτάνουν στη χώρα, στη χώρα του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι λοιπόν σε κάποιες χώρες μέλη η κατάσταση αυτή ελέγχεται, ρυθμίζεται αυστηρά, σε άλλες λιγότερο. Σε κάποιες χώρες έχουμε υψηλή ζήτηση, σε άλλες χώρες λιγότερη ζήτηση. Ε, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο εθνικός προστατευτισμός πολύ συχνά δεν είναι ένας προστατευτισμός εθνικιστικού χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι προκαλείται περισσότερο από τις επαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες ασκούν ε, πίεση στην εσωτερική αγορά εργασίας της κάθε χώρας. Για να συμβάλλω θετικά σας κάνω μια πρόταση. Νομίζω ότι οι μελέτες που θα κάνει η Επιτροπή σε αυτό το τομέα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τις ιδιάζουσες ε, καταστάσεις στην αγορά εργασίας στην κάθε χώρα μέλος επειδή υπάρχουν και άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΑΣΑ ο οποίος ήδη δημοσιεύει στοιχεία για το κόστος της επαγγελματικής ε, της συνομιατρικής επίσκεψης στις χώρες του ΟΣΑ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσα θα ήταν δυνατόν να το κάνουμε αλλά νομίζω ότι δεν έχει πια νόημα να κάνουμε συγκρίσεις όσον αφορά την μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών εάν δεν κάνουμε το απαραίτητο, δηλαδή να δούμε τι γίνεται στην εσωτερική αγορά της κάθε χώρας, κατά πόσο υπάρχουν επαγγελματικοί φραγμοί, νομοθετικοί φραγμοί κλπ. κλπ. Ευχαριστώ. Oui, Να έχετε δίκιο. Για να... Α, όχι, συγγνώμη, σας ξέχασα. Κόντεψα να ξεχάσω τον ε, συνάδελφο. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Μπερναντέτ, που μου ξαναδίνει το λόγο. Θα ήθελα να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα στους εμπειρογνώμονε Για τα ιατρικά επαγγελματά όλοι μιλούν για τον ιατρικό κίνδυνο. Η ερώτησή μου είναι απλή. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να, ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε επειδή δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Αλλά τα στοιχεία αυτά είναι σωστά. Αν θα υπήρχαν. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το επιχείρημα βεβαίως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για να τεθούν φραγμοί. Στην Γαλλία θεωρούμε κάθε χρόνο ότι 10 με 50.000 10, με 50.000 ε, ασθενείς πεθαίνουν στα γαλλικά νοσοκομεία από περιπλοκές που οφείλονται στην ιατρική δραστηριότητα, ή από ιούς νοσοκομιακούς ή από έλλειψη σωστής γνώσης της γλώσσας κλπ. κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτό τον τεράστιο ρυθμό ασθενών που πεθαίνουν κάθε χρόνο και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το θέμα των ιατρών που είτε έχουν λάβει κακή εκπαίδευση είτε έχουν πάει να εργαστούν παράνομα σε κάποια χώρα δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι αυτά τα άτομα λοιπόν βρίσκονται στο ύψο των περιστάσεων. Δηλαδή θέλω να πω ότι στατιστικά το πρόβλημα νομίζω ότι είναι τεχνητό. Μήπως λοιπόν αυτό που λέγαμε προηγουμένω αποτελεί ένα άλοθη για τον παρεμποδισμό στη δικασία τη ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ θα προσθέσω ένα στοιχείο το οποίο σκέφτηκα τώρα μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφος Ζιβά, δηλαδή η οδηγία για τα ιατρικά επαγγέλματα που αφορούσε την διασυνοριακή περίθαλψη. Σε μια ομάδα εργασίας είπαμε ότι δεν χρειάζεται να προβλέπουμε τον ιατρικό κίνδυνο επειδή αυτό είναι ελάχιστο ή αμεληταίος. Είχαμε λοιπόν πολύ γενικόλογα, γενικά και όλες τα στοιχεία και νομίζω ότι για τον ιατρικό κίνδυνο οι στατιστικές είναι αυτές που είναι αλλά ήδη σήμερα ενδεχομένω από την συζήτησή μας μπορεί να ανακύψει κάτι θετικό σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ο λόγο στον κύριο Φορτούι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που τέθηκαν από το σύνολο των βουλευτών πριν από λίγο. Είναι δύσκολο να τα συνοψίσει κανείς. Καταρχήν θα μιλήσω ως φαρμακοποιός επειδή η αποστολή μου ήταν κάτι το οποίο σχετιζόταν με τους φαρμακοποιούς. Είχα οριστεί και εμψυχωτής σε μια ομάδα στην Asprocard που ανταποκρίνεται στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και που τους αφορούσε άμεσα η οδηγία. Μιλάμε για τους φαρμακοποιούς, νοσοκόμους, οδοντιάτρους ε, χειρουργούς κλπ. κλπ. Είναι σαφές ότι για αυτή την αποστολή και γι' αυτό ακριβώς ε, λαμβάνω το θάρρος να πω δύο λόγια. Γι' αυτή την αποστολή λοιπόν μετακινηθήκαμε, συναντήσαμε όλες τις αρμόδιες αρχές των ευρωπαϊκών χωρών και όπως σας έλεγα προηγουμένως έχουμε να κάνουμε με τους ε, επαγγελματίες του ιατρικού χώρου συναντήσαμε και υπαλλήλου από Υπουργεία και άλλους φορείς και μπορώ να σας πω ότι υπήρξε αντίθεση τοπικά ενδεχομένω, αλλά νομίζω ότι σφαιρικά δεν υπήρξε αντίθεση ή διχογνωμία μεταξύ του Γαλλικού Υπουργείου Υγείας και των φαρμακοποιών ας πούμε. Εγώ ως φαρμακοποιός προσπαθώ να μην έχω περιορισμένη οπτική γωνία, δηλαδή κάτι το οποίο να άπτεται του προστατευτισμού όσον αφορά ας πούμε, την άφηξη φαρμακοποιών από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γαλλία. Δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα που ανέφερα προηγουμένω, επειδή θέλαμε ακριβώ να διευκολύνουμε την κινητικότητα, τι προποθέσει και του όρου τη κινητικότητα, το οποίο είναι διαφορετικό από την κινητικότητα αυτή καθεαυτή. Πρέπει να σημειώσουμε και να καταγράψουμε αυτή τη διαφορά. Βεβαίω, έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια των ασθενών εδώ, αλλά όπως είπατε και εσείς δεν έχουμε στοιχεία στη διάθεσή μας. Δεν γνωρίζουμε, κανείς δεν γνωρίζει και επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσους ε, έχουμε στην Ευρώπη που ασχολούνται με τα ιατρικά επαγγέλματα. Να δούμε τα στοιχεία από τις μελέτες συλλέγοντα στοιχεία από τι αρμόδιε αρχέ ή καταλόγου επαγγελματικού, τότε θα δούμε ότι υπάρχουν σημαντικέ αποκλήσει όσον αφορά το σύνολο των επαγγελματιών αυτών. Συναντήσαμε τους υπεύθυνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και κοιτάξαμε να κάνουμε κάτι από κοινού όσον αφορά τους επαγγελματίες του ιατρικού χώρου. Άλλοι λαμβάνουν υπόψη του στο σύνολο των εργαζομένων, άλλοι μόνο κάποιες ειδικότητε ή κάποια επαγγέλματα, άλλοι λαμβάνουν ας πούμε τα στοιχεία που αφορούν τους ασθενείς και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα στοιχεία αυτά δεν είναι σαφή, δεν είναι πλήρη. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι αξιόπιστα αυτά τα στοιχεία. Σήμερα λοιπόν υπάρχει πράγματι κάποια οριστία για τα στοιχεία που λέγαμε, οπότε εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη διορθώσουμε. Προηγουμένως αναφέρθηκα στις ευρωπαϊκές δομές και στη αρμοδίων αρχών που θα θέλαμε να υλοποιήσουμε. Αυτό ήταν και η τελευταία απόφαση της ομάδας εργασίας να δούμε δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε, να συγκαλέσουμε τις αρμόδιες αρχές. Και ξέρετε όταν κάναμε τον απολογισμό είδαμε ότι στην Ευρώπη είχαμε 890 αρμόδιες αρχές για τα πέντε λόγω επαγγέλματα. 890. Αν λάβω υπόψη μου α πούμε την Εστονία. Η Εστονία έχει μια αρχή αλλά δεν έχει καμιά αρχή και για τα πέντε επάγγελματα. Στη Γαλλία, α πούμε, έχουμε πέντε διαφορετικέ αρχέ, μία ένα επάγγελμα. Στην Ιταλία, δεν έχω τίποτα εναντίον τη Ιταλία βεβαίω. Ε. άλλο γιατί συνεργαστήκαμε πολύ με του Ιταλού που ήδη για τους ε, ιατρούς έχουν μια κάρτα επαγγελματική ευρωπαϊκή. Για την Ιταλία έχουμε λοιπόν αρμόδια αρχή επαγγελματική αναπεριφέρεια. περιφέρεια. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική δουλειά συντονισμού που θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε και εδώ ακριβώς θα μπορούσε να γίνει μια ενδιαφέρουσα δουλειά μεταξύ των ευρωβουλευτών, των αρμοδίων αρχών που είμαστε εμείς και των επαγγελματικών οργανώσεων. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματική οργάνωση, αποτελούμε ένα είδος ε, τάγματος αν θέλετε Έχουμε διαφορετική επαγγελματική διοντολογία, δεν ακολουθούμε ε, οικονομικές προσταγές, δεν είναι αυτή η βούλησή μας, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά σε συνεργασία όλοι μας και μαζί με τις αρμόδιες αρχές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, είμαι βεβαία και το εύχομαι τουλάχιστον ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυνεργαστούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χέιζελ, τον άλλο εμπειρογνώμονα, να απαντήσει κι αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι δύσκολο βέβαια να εκπροσωπήσω τις 27 αρμόδιες αρχές ε, για τις ΜΕΣ. Θα περιοριστώ στο Εθνικό μας Συμβούλιο. Το θέμα του ιατρικού κινδύνου είναι ενδιαφέρον. Το Ιατρικό Συμβούλιο έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία πάνω σε αυτό και θυμάμαι ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου ανέφερε κάποια στιγμή ότι οι ξένοι γιατροί που έχουν πτυχία ε, από το εξωτερικό, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ε, έχουν διπλάσια πιθανότητα να εμφανιστούν μπροστά σε κάποια κροαματική διαδικασία για την πρακτική τους. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ακριβές απόλυτα βέβαια. Επίσης ε, τα πρότυπα πρόσφατα Έχουμε θεσπίσει νέα πρότυπα για την εκπαίδευση των νοσηλευτών. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και το ε, αποτέλεσμα όλων αυτών. Είναι σημαντικό να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, για την εκπαίδευση έχουμε ε, ένα φορέα παροχής γνώσεων που είναι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και είναι και επιγραμμική η εκπαίδευση, ιδιαίτερα η θεωρητική βέβαια με εκπαιδευτικές κλίμακες, αλλά δεν υποκαθιστά αυτό την πρακτική εκπαίδευση που χρειάζονται οι νοσηλευτές και οι ΜΕΣ. Πολλοί όμως εκμεταλλεύονται τις ε, ευκαιρίες αυτές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τώρα, ε, Πώς όλα αυτά επηρέασαν τη διακίνηση των εργαζομένων. Ήταν πολύ θετική η επίπτωση όλων αυτών, αυξήθηκε η κινητικότητα και αναγνωρίζουμε και την ε, συμβολή αλλοδαπών, μεών και νοσηλευτών. Εμείς έχουμε περίπου 7.000 αιτήσει από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο στα πλαίσια της οδηγίας. Ένα θετικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι το ε, δίκτυο που δημιουργήσαμε θα συνεχιστεί. Εμείς έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να συνεργαστούμε και Χαίρομαι που θα συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των 27 αρμοδίων αρχών και θα υπάρχει ευκαιρία να μοιραστούν ε, γνώσεις, να επικοινωνήσουν περισσότερο και να συνεργαστούν για να είναι πιο τυποποιημένες οι διαδικασίες. Τώρα για την επαγγελματική κάρτα και εδώ ο φορέας μας ήταν πολύ δραστήριος και συμμετείχαμε σε συζητήσεις. Είδαμε όμως ε, κάποια πρακτικά προβλήματα. Δεν είμαστε ε, καταρχήν κατά, αλλά όπως είπα και πριν έχουμε περίπου 650.000 μέλη στο μητρό μας. Ορισμένοι εργάζονται στα βρετανικά νησιά και σε υπερπόντιες περιοχές, Γιβραλτάρ, Φόκλαντ κλπ. Και έχουμε και 10.000 που εργάζονται στο στρατό, σε ένοπλες δυνάμεις. Οπότε υπάρχει θέμα logistics στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπέρ της αντίληψης αυτής και αν χρησιμοποιηθεί θετικά και επικοδομητικά, σίγουρα μας ενδιαφέρει να το εξετάσουμε και πάλι πιο προσεκτικά. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν μου ξέφυγε καμία, ευχαρίστω να επανέλθω και να απαντήσω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα πέντε λεπτά πριν από την άφηξη του κυρίου Μπαρνιέ. Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις αυθόρμητες που ανέκυψαν. Έχω μία, αν δεν υπάρχουν άλλες, λέει πρόεδρος. Θα τη θέσω στους εμπειρογνώμονες, γιατί μιλήσαμε πολύ για την γλωσσική κατάρτιση και την ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση των επαγγελματιών που μετακινούνται ιδιαίτερα στα ιατρικά επαγγέλματα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών αλλά και η ασφάλεια η νομοθετική των επαγγελματιών Αναστησιολόγοι, χειρούργοι, όλοι αυτοί πρέπει να σε να επικοινωνούν τους ασθενείς αν έχουν κάποια αλλεργία κλπ. Αυτή λοιπόν η επαγγελματική κάρτα θα μπορούσε να ήταν υποχρεωτική στην χώρα υποδοχής. Η, η ταχεία γλωσσική κατάρτιση τριών εβδομάδων επαρκεί ή θα πρέπει να γίνεται μια περισσότερο εις βάθος εκπαίδευση για αυτά τα θέματα. Ποια είναι η απόψη σας. Όποιος από τους δύο θέλει να γινεται μια περισσοτερο εις εκπαιδευση για αυτα έχουμε χρόνο. Για την χρήση της γλώσσας υποδοχής πραγματικά αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ξέρετε ότι όπως λέμε σε εισαγωγικά συνίσταται έντονα να μην προσλαμβάνουμε επαγγελματίες που δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση εκπαίδευση ή γλωσσική εκπαίδευση. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε βέβαιοι ότι ο Τάδιο Δίνα επαγγελματία που κατάγεται από άλλη χώρα μιλάει καλά τη γλώσσα, τότε εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν κάποιος Βέλγος έρχεται στη Γαλλία θεωρούμε ότι μιλούν γαλλικά. Όταν όμως έχουμε αμφιβολίες για μια χώρα ή για κάποιον που έρχεται από μια πιο μακρινή χώρα, τότε παίρνουμε το τηλέφωνο με πρόσχημα τέλο πάντων τη ε, συμπλήρωση κάποιων στοιχείων του φακέλου του και του μιλάμε. Να δούμε ακριβώ τι γνώσει έχει. Σήμερα πάντω δεν έχουμε το δικαίωμα να του θέσουμε το ερώτημα άμεσα και κατά κάποιο τρόπο να τον ανακρίνουμε. Αυτό λοιπόν ενδεχομένω δεν φαίνεται σωστό και δεν νομίζω να βοηθάει την ασφάλεια των ε, ασθενών. Ε, επ' αυτού θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Όπως είπα στην παρουσίαση, οι περισσότερες αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν ότι το θέμα της γλώσσας ήταν κυρίαρχο για τους εργοδότες και η Βαρόνη παρουσίασε σωστά τον ρόλο του, της ρυθμιστικής αρχής σε αυτά τα θέματα και είπε ότι υπάρχουν θέματα όμως που θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Θα ήθελα να κάνω μια διάκριση εδώ σε αυτό το πλαίσιο η καταλληλότητα για άσκηση επαγγέλματο και η καταλληλότητα για γραφή στο Μητρό δεν είναι το ίδιο. Είναι ξεκάθαρο ότι η έλλειψη γλωσσικής δεξιότητας αποτελεί ένα σημαντικό θέμα τουλάχιστον στο 50% των θεμάτων που έθιξαν οι αρμόδιες αρχές για τις ΜΕΕΣ και τις νοσοκόμες. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε νομίζω με δεξιότητες επικοινωνίας και αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και αυτοί που εκπαιδεύονται στην χώρα τους, αλλά και αυτοί που μετακινούνται. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποεκτιμάμε την δεξιότητα για κατάλληλη επικοινωνία σε οποιοδήποτε τομέα επαγγελματικό και υπό οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Θέλετε εσείς κυρία μου να προσθέσετε κάτι? Όχι. Ναι, αρνητικά. Όχι. Κύριε Ζουβά, έχω δύο αγορητές που ζητούν το λόγο, ο κύριος Φεσνερ και ο κύριος Ζουβά. Θυμήθηκα το εξής. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις επίσης, ας πούμε Βρετανών πολιτών, που περνούν πολύ χρόνο στην Ισπανία γιατί ένας μη ισπανόφωνος Βρετανός γιατρός να μην εγκατασταθεί και να ασκήσει το επάγγελμά του εκεί. Και αυτό πρέπει να απασχολήσει την ε, αγορά. Και ενδιαφέρει την αγορά. Γιατί θα ενδιαφέρει και άλλους που βρίσκονται εκεί. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό, αλλά κάποιο μπορεί να ενδιαφέρεται να εξυπηρετηθεί από ένα Βρετανό που είναι στην Ισπανία να πάει σε έναν Ισπανό γιατρό. Ε, και δεν καταλάβαινα κι εγώ. Έχω πάει πολλέ φορέ στην Ισπανία, δεν καταλαβαίνω πώ δεν μιλάνε ούτε μία, γλω... ούτε μία λέξη αγγλικά, ή, συγγνώμη, ισπανικά, οι Άγγλοι που ζουν στην Ισπανία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι, κατανοούμε, λέει ο κύριο Ζιβάν πόσο περίπλοκο μπορεί να είναι το θέμα, λοιπόν. Ε, συμφωνώ απολύτω άλλωστε με αυτό αυτά που είπε. Ε, υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιες, ε, κάποια επαγγέλματα που δεν είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς τη γλώσσα καλά. Όταν δηλαδή ε, κανείς ε, προσλαμβάνεται για μια θέση η οποία δεν έχει επαφή με το κοινό, με τους πελάτες που ε, χρειάζεται απλώς ε, να έχει κάποιες τεχνικές γνώσεις. Προφανώς δεν υπάρχει λόγος, αλλά υπάρχουν, ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπως ας πούμε και ο φαρμακοποιός που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και οπωσδήποτε πρέπει να ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα. Η η μη δυνατότητα επιβεβαίωσης του επίπεδου γνώσης της γλώσσας δημιουργεί πρόβλημα και για την πλευρά του παρουσιαζόμενου ε, επαγγελματία αλλά και ε, τον, ε, από την πλευρά αυτού που πρόκειται να τον προσλάβει. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι είναι πλέον, δεν είναι πλέον νόμιμο, επομένως είναι παράνομο το να ανακρίνει κανείς ε, κάποιον για να ξέρει ή να καταλάβει αν γνωρίζει τη γλώσσα ή όχι αλλά και ο ίδιος δεν μπορεί να υποβάλει παραπάνω παραστατικά από αυτά ε, τα οποία ε, ζητώνται. Ε, βεβαίως μπορεί να εφεσιβάλει κάποια απόφαση λέγοντας ότι εγώ έχω έξτρα γνώσεις, επιπλέον γνώσεις που είναι αυτά τα διπλώματα κτλ. Εφαρμόζουμε, εφαρμόζουμε λοιπόν έναν κανόνα ο οποίος υποτίθεται ότι δεν υπάρχει. Τον εφαρμόζουμε και εσφαλμένα και μετά δεν μπορούμε καν να προσφύγουμε κατά της απόφασης που απορρέει από την ασφαλμένη χρήση. Ο κύριος Αντρός Παλέρ από την ε, Ουγγαρία έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Ρέπο, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη συζήτηση περιμένοντας τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συνεδρίαση όπου ακούσαμε πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις. Ελπίζω να ξανασυνεδριάσουμε τους επόμενους έξι μήνες υπό Ουγγρική Προεδρία. Δύο πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω. Αν γίνεται, νομίζω θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε την οδηγία αυτή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται νέες αρμοδιότητες. Μιλήσαμε για έκδοση πτυχίων από διάφορες αρχές, μιλήσαμε για συνεργασία αρχών, μιλήσαμε για πλαίσια, μιλήσαμε για το κατά πόσο ένα πτυχίο είναι γνήσιο ή όχι. Ωραία όλα αυτά. Διερωτώ με, ως πολίτης που μιλάει μια γλώσσα τελείως διαφορετική από αυτή των υπολείπων πολιτών της Ευρώπης, κατά πόσο το θέμα της γνώσης της γλώσσας πώς θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με το όλο θέμα της εκπαίδευσης. Δηλαδή θα έπρεπε να δούμε ακριβώς το επίπεδο των διαφόρων γλωσσικών κύκλων μάθησης και ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε αν τα κριτήρια που θα έπρεπε να εφαρμόσουμε εδώ στο, στο θέμα της γλώσσας θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να εναρμονιστούν. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, πολύ, καλό, πολύ καλή παρατήρηση. Ο κύριος Τρεπό θα θέσει ένα ερώτημα ή κάποιο συμπέρασμα, δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ μιλάω φιλανδικά, μια εξίσου σπάνια γλώσσα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και ιδιαίτερα για τα σχόλια που έκανε ο συνάδελφος γιατρός προηγουμένως, τα οποία ήταν πολύ ευφυή. Αλλά ως απλός άνθρωπος θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό της γλώσσας στον τομέα των ιατρικών επαγγελμάτων είναι κατά κάποιο τρόπο αναλογικό. Δηλαδή στη Φιλανδία μια από τις κυριότερες ειδήσει φέτος το καλοκαίρι ήταν ότι είχαμε έναν ψευτογιατρό που ασκούσε το επάγγελμα για δύο χρόνια χωρίς καμία κατάρτιση και πώς, δινόταν, πώς γινόταν αυτό γινόταν επειδή ήταν πολύ καλός στις γλώσσες. Δηλαδή ζητούσε συμβουλές για κάθε νόσο όλους τους συναδέλφους. Είχε λοιπόν πολλά στοιχεία και πολλές πληροφορίες επειδή μιλούσε πολύ καλά τη γλώσσα. Η γλώσσα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά εδώ βεβαίω θα μπορούσε να δημιουργήσει και προβλήματα όπως βλέπετε. Ευχαριστώ. Ε, οι συνάδελφοι προσθέτουν προβλήματα εκεί που πραγματικά καμιά φορά δεν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποδεχτώ τον Επίτροπο τον κύριο Μπαρνιέ και να του πω ότι με χαρά τον υποδεχόμαστε εδώ στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς όπου για σύντομο χρονικό διάστημα ήταν συνάδελφός μας γνωρίζει πολύ καλά την κοινοβουλευτική διαδικασία γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όπως το έχω ξαναπεί είναι ένας από τους λίγους επιτρόπους που έχει μια ευρωπαϊκή οπτική Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ας είμαστε ειλικρινείς, έτσι είναι. Ελάχιστοι έχουν ευρωπαϊκή οπτική και αντιμετωπίζουν την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Μπαρνιέ και να συγχαρώ εσά και τις υπηρεσίες σας γιατί την περασμένη Παρασκευή εκδώσατε τα συμπεράσματα της έκθεσης για τη μεταφορά της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητε. Ξέρω ότι αυτή η εργασία ήταν τεράστια που έκαναν οι υπηρεσίε σα. Εξώματο λοιπόν τη Επιτροπή Ενιαία αγορά και όλους, όλα τα, τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία ευχαριστώ για την παρουσία του. Σα ευχαριστούμε. Ξέρω ότι είχατε σημαντική δουλειά να κάνετε γιατί είχαμε μια προδημοσίευση στο ΕΚΟ χθες για την αυριανή ανακοίνωση που θα κάνετε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ σήμερα. Ξέρουμε ότι έχετε πολλή δουλειά. Θα σας δώσω το λόγο. Γιατί ξέρω ότι έχετε πολλά θέματα να θίξετε. Έχουν μείνει πολλά θέματα ακόμα που θα πρέπει να διευκρινιστούν, αλλά είμαστε στον καλό δρόμο γιατί έχουμε την πολιτική βούληση, η οποία προέρχεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε τα τρία θεσμικά όργανα τη Ένωση, να συνεργαστούν μαζί με του αδέλφου των 27 χωρών που εκπροσωπούνται από τα Εθνικά Κοινοβούλια σας δίνω λοιπόν το λόγο για μισή ώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν οπωσδήποτε ευρωπαϊκό όραμα. Ενδεχομένως ε, βλέπουν ε, το θέμα από διαφορετική γωνία, έχουν διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας, αλλά παρόλα αυτά Νομίζω ότι σε αυτό το κολέγιο των επιτρόπων επικεφαλής του οποίου είναι ο πρόεδρος Μπαρόζο υπάρχει μια σαφής ευρωπαϊκή προοπτική. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτέ που βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας. Δυστυχώς πρέπει να φύγω γρήγορα μετά από την παρέμβασή μου, γιατί όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, αύριο μαζί με 12 συναδέλφους θα υποβάλω μία πρωτότυπη εργασία την οποία ονομάσαμε Single Market Act, πράξη ε, για την ενιαία αγορά. Μια νέα διάσταση της ε, ε, ενιαίας αγοράς ε, που θα αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα είναι φτιαγμένη για αυτές και θα αφορά τους καταναλωτές και τους πολίτες και θα είναι φτιαγμένη για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει αγαπητοί φίλοι να ψάξουμε την ανάπτυξη εκεί που ακριβώς υπάρχει. Έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών που επομένως εάν λειτουργήσει η αγορά αυτή καλύτερα από ό,τι λειτουργεί σήμερα δυνητικά μπορεί να έχουμε πάρα πολύ καλή ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δημιουργήσουμε αγορά χωρίς τις εταιρείε ή ενάντια στις εταιρείε, χωρίς τους πολίτες ή ενάντια στους πολίτες. Πρέπει όλοι μαζί λοιπόν ε, να κινηθούμε. Ε, βεβαίως θα ήθελα να χαιρετήσω και τους ε, Ευρωπαίους βουλευτές. Ήμουν κάθισα στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αλλά έχω καθίσει και στα έδρανα του Εθνικού μου Κοινοβουλίου και επομένως δεν ξεχνώ ποτέ ε, αυτήν την ε, εμπειρία μου και νομίζω ότι στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πρέπει να προσπαθούμε να συνδέουμε την συζήτηση του σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την συζήτηση σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτήν την μεγάλη εσωτερική αγορά των πολιτών. Αύριο μάλιστα στην παρουσίαση της ε, ε, έκθεσής μου ε, θα αναφερθώ σε όλα τα θέματα αυτά και η έκθεση της κυρίας Γκρέσ μάλιστα πολλά στοιχεία περιλαμβάνει ε, τα οποία θα ακουστούν ε, αύριο και μην ξεχνάμε και βεβαίως το βάρος και τη σημασία του έργου αυτής της ομάδας εργασίας που δημιουργήσετε για τα επαγγελματικά προσόντα. παρακολουθούμε όλες αυτές τις κινήσεις με πάλι πολύ μεγάλη προσοχή. Θα σας μιλήσω άμεσα και ειλικρινά για το θέμα ε, αυτό το οποίο αφορά την ανθρώπινη διάσταση αυτής της μεγάλης ενιαίας αγοράς. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία μεγάλα σημεία. Τι κάναμε όσον αφορά την οδηγία αυτή. Δεύτερον, που βρισκόμαστε σήμερα. Και τρίτον, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να πάμε εμπρός, να προχωρήσουμε, να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Και ποια είναι βεβαίως και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο μου είχατε υποβάλει ένα προφορικό ερώτημα και το οποίο είχαν προσυπογράψει πολλοί βουλευτές Πρέπει να πω ότι τότε βέβαια δεν ήμουν ακόμα επισήμως, δεν είχα επισήμως αναλάβει την θέση μου και τις αρμοδιότητες που έχω τώρα ως επίτροπος, αλλά ε, εξέφραζαν ε, την ε, ανησυχία τους και την ανεκανοποίησή τους πολλοί βουλευτές όσον αφορά την ενσωμάτωση της οδηγίας. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευτυχή και σίγουρα ανακοφισμένο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωση σε όλε τι χώρε μέλη και, στα, και στι 27 χώρε δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά, δεν κατανοώ, δυσκολεύομαι λοιπόν να καταλάβω γιατί χρειάστηκε, να, χρειάστηκε τόσους χρόνους, τρία χρόνια για να μεταφερθεί αυτή η οδηγία. Η οδηγία αυτή λοιπόν έγινε δεκτή το 2005 και ε, στην ουσία επιβεβαίωνε παλαιότερα ή υφιστάμενα κείμενα. Και αναρωτιέμαι με έκπληξη γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος έτσι ώστε να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Ενώ ήδη οι περισσότερες διατάξεις είχαν ήδη ενσωματωθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι δεν ήταν προτεραιότητα για αυτά. Ίσως. Εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν 4.600 ε, επαγγέλματα ρυθμισμένα, 4.600. Γι' αυτό λοιπόν με τόσες ε, με τόσα επαγγέλματα ρυθμισμένα που εκπροσωπώνται και σήμερα εδώ και χαιρετίζω τους εκπροσώπους τους. Ίσως το πράγμα έγινε πολύ περίπλοκο από τους γιατρούς μέχρι τους ε, αρχιτέκτονες, από τους ε, μηχανικούς ε, μέχρι τους δάσκαλους του, δασκάλου, συγγνώμη, του σκι μιλάμε για την καθημερινότητα πολλών Ευρωπαίων επαγγελματιών ή πολλών πολιτών που, στους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους αυτοί οι επαγγελματίες. Αυτό όσον αφορά την ασωμάτωση της οδηγίας. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ε, στην υφιστάμενη διαδικασία αξιολόγησης. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία κινητοποιεί πολύ κόσμο εμείς ξεκινήσαμε τον προηγούμενο Μάρτιο τη διαδικασία αξιολόγησης οδηγίας προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον ε, και από τα κράτη-μέλη που συμμετέσχουν σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Πολύ μεταξύ ημών κυρίες και κύριοι επιστήσατε την προσοχή μας στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με το κείμενο και την ε, εφαρμογή του. 25 γραπτές ε, και προφορικές ερωτήσεις δέχτηκα από μέλη του Κοινοβουλίου και εγώ ο ίδιος ε, που γνωρίζετε ίσως ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μια πρωτεύουσα ε, έχω, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην ε, Πολωνία, έχω πάει στην Πορτογαλία, στην Ουγγαρία, στην Πορτογαλία, στην Αυστρία Κάθε εβδομάδα λοιπόν πηγαίνω κάπου σε μια πρωτεύουσα ε, και δημιουργώ ένα workshop, μια ομάδα εργασίας για την ε, εσωτερική αγορά με όλους τους εμπλεκόμενους ε, φορείς και εκεί αναφέρεται πάντα και η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα ενώπιον της πολωνικής διέτης και σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσω μαζί σας. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πέρα από τις ε, πολλές ερωτήσεις που έχουν ε, υποβάλει οι Ευρωπαίοι βουλευτές έχω και τα, τις ερωτήσεις των εθνικών βουλευτών. Επίσης έχουμε οργανώσει και ακροάσεις με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών των διαφόρων κλάδων και φορέων. Ξέρω ότι ακούσατε τον κύριο Φορτουή πριν από λίγο, τον κύριο Χέιζελ ε, που εκπροσωπούν, ε, τους χαιρετίζω μάλιστα γιατί βλέπω ότι είναι εδώ ε, και που σας μίλησαν για τα προβλήματα κάποιων επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα ε, και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα το, μετά το πέρας των αξιολογήσεων όλων των επαγγελματικών φορέων δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα των ερευνών την 21η Οκτωβρίου γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Περάσαμε λοιπόν από το πρώτο στάδιο που ήταν η μεγάλη διαβούλευση ε, και όλη η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Εγώ θα προσπαθήσω μαζί σας ε, να ε, εξαρτηθώ κάποια πρώτα συμπεράσματα, κάποιες οδούς βελτίωσης. Τρεις είναι οι κύριες οδοί. Μια μεγαλύτερη απλούστευση πρώτον εξυγχρονισμός του κεκτημένου των προσόντων και περισσότερη proactive συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Μεγαλύτερη απλούστευση σας είπα. Οι διαδικασίες στα κράτη-μέλη πολύ συχνά είναι μακροσκελής, είναι γραφειοκρατικές, αδιαφανείς, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων με συνεχή τρόπο ε, αντιπροσωπεύει το 20% ε, του δικτύου Solvit. Στην Βασοβία ξέρω ότι η ομάδα Solvit λειτουργεί πάρα πολύ καλά. 20% λοιπόν των υποθέσεων που φτάνουν στη Σολβίτ αφορούν την ε, γραφειοκρατική βραδύτητα, την μη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων κλπ. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα περαιτέρω απλούστευσης, κυρίως για να βελτιώσουμε, ε, κυρίως όσον αφορά μάλλον την προσωρινή κινητικότητα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να βελτιώσει την προσωρινή κινητικότητα και τώρα τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να ζητήσουν από τον ενδιαφερόμενο ε, εργαζόμενο, ο οποίος ενδιαφέρεται δηλαδή για προσωρινή κινητικότητα, ε, να υποβάλουν μία ε, πρώτερη δήλωση. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις από πλευράς των κρατών. Έχουν τα κράτη βαρύνει πάρα πολύ τη διαδικασία με τρόπον ώστε και σε σημείο ώστε να απογυμνώσουν τελείως τελικά τις δυνατότητες που αρχικά εδίδονται μέσω των διατάξεων για την προσωρινή κινητικότητα. Επίσης ε, ε, σε πολλές ε, περιπτώσεις ζητώνται ας πούμε τα πρωτότυπα και μάλιστα επικυρωμένα των διπλωμάτων πράγμα που σημαίνει ότι έρεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα υποβολής επιγραμμικά των όποιων πιστοποιητικών. Εμείς θέλουμε και το λέμε στην Single Market Act να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι ηλεκτρονικές δυνατότητες. Δεύτερο, θα θέλαμε να βελτιώσουμε το κεκτημένο όσον αφορά την αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων αρχιτέκτονες. Αυτό που έγινε εκεί νομίζω ήταν επιτυχία και συμφωνείτε κι εσείς ότι το, επειδή το σύστημα αυτό όχι μόνο έγινε αποδεκτό από τους επαγγελματίε που ενδιαφέρει άμεση αναγνώριση αλλά και από την μεγάλη πλειοψηφία αρμόδιων αρχών είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια άμεση αναγνώριση που είχε αρχικά εφαρμοστεί για 6 χώρες είναι διαθέσιμη στις 26. Βεβαίως μετά από την θέσπιση του συστήματος θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ενημερώσουμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης που πολλές φορές ανάγονται σε δεκαετίες στο παρελθόν περίπλοκο αυτό, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αρχή τη αμοιβαία και αυτόματη αναγνώριση θα πρέπει να διατηρηθεί. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελμάτων, η αναγνώριση των πτυχίων δεν είναι, δεν είναι αυτόματη, αλλά βασίζεται σε αναγνωρίσει αναπερίπτωση πώς θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε πτυχία τα οποία έχουν ληφθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα όσον έχουμε να κάνουμε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορες χώρες και μάλιστα είχαμε και τη διαδικασία της Μπολόνια για τα πανεπιστήμια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν μια σημαντική μελέτη εις βάθος για να εξετάσουμε το πώς ακριβώς οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αναγνώριση των πτυχίων. Τρίτο σημείο είναι η ενεργητική συνεργασία. Πρόεδρε, έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα από ευρωβουλευτές και αφορούν ιατρούς οι οποίοι ασκούν παράνομα το επάγγελμά τους. Αυτοί μπορούν να απολαύσουν τις ελεύθερες μετακίνησης. Όχι. Έχαμε την περίπτωση ενός γιατρού που δεν μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμά του στην Ισπανία και το έκανε στη Βρετανία. Αυτό το θέμα έκανε να χυθεί πολύ μελάνη πρόσφατα, κάτι το οποίο μας καταδεικνύει ακριβώς την ανάγκη προώθησης μιας συνεργασίας ενεργούς μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών βεβαίως και ιδιαίτερα των αρχών που αφορούν τους ε, ανθρώπους που εργάζονται στα ιατρικά επαγγέλματα. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Βεβαίω, όλη αυτή η διαπίστωση, όλε αυτέ τι διαπιστώσει που έκανα τηλεγραφικά μα προσφέρουν κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι θα πρέπει δηλαδή να πάμε σε μια εξυγχρόνηση της οδηγίας και θα ήθελα να σας πω ότι έχω πρόθεση το φθινόπωρο του 2011 να παρουσιάσω ένα, μια πράσινη βίβλο και το 2012 μια νομοθετική πράξη Προ την κατεύθυνση αυτή. Θα εξετάσουμε βεβαίω τι διάφορες προβληματικές που έχουν ανακύψει όσον αφορά τι ε, αξιολογήσει ή κατά διάρκεια των αξιολογήσεων και επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που θα έρθουν στην Επιτροπή από την Ευρωβουλή, τα Εθνικά Κοινοβούλια, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους μεμονωμένους πολίτες και θα ήθελα να σας πω για αυτό το θέμα ότι διαβουλεύσεις που θα ξεκινήσουμε από αύριο από το Synchron Market Act μια δημόσια συζήτηση. Αυτή την πράξη για την νέα αγορά θα την στείλω σε κάθε βουλευτή της Ευρώπης θα μεταφραστεί σε 23 γλώσσες για να διευκολύνουμε τη συζήτηση και στις περιφέρειες θα σταλεί και εγώ πραγματικά θα δώσω ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που θα ανακύψουν από τη δημόσια συζήτηση. Θα είμαι λοιπόν ευήκο ό,τι λάβω ω παρατηρήσει και σχόλια από βουλευτέ, επαγγελματικέ οργανώσει κλπ. Και έχω ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τι προσδοκίε των ασθενών και των καταναλωτών, γιατί η κινητικότητα των ιατρικών επαγγελμάτων και οι ενσυχίες που ακούστηκαν σε σχέση με αυτό το θέμα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την γλωσσική επάρκεια όσον αφορά την άσκηση ενός επαγγέλματο και επιθυμίσω ότι σύμφωνα με την οδηγία πρέπει κανείς να έχει γλωσσική επάρκεια για να ασκήσει το επάγγελμά του. Οι χώρες μέλη μπορούν να το ελέξουν αυτό και επ' αυτού αναμένουμε οι χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν ακριβώς και να ασκήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τωρινή οδηγία. Ένα δεύτερο σχόλιο για το θέμα αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι η οδηγία δεν αποβλέπει μόνο στον τομέα της υγείας στα ιατρικά επαγγέλματα. Περιλαμβάνει και άλλα επαγγέλματα που αφορούν εκατομμύρια πολίτες που ασκούν επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες ε, επαγγελματίες που υποβάλλουν αίτηση αναγνώριση σε άλλη χώρα και πολλούς άλλους ε, τους οποίους ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό ατόμων που μετακινούνται προσωρινά και γι' αυτό κυρίε και κύριοι πρόκειται για μια οδηγία κλειδί για τους πολίτες αλλά και για τις αγορές μας αλλά και για την οικονομία μας. Το αίτημα των εργαζομένων, μάλλον το, η, ζήτηση, η ζήτηση για εργαζόμενους με υψηλή κατάρτιση θα αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι γύρω στα 16 εκατομμύρια ο αριθμός αυτός και είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτή η ζήτηση από το τωρινό τον υπάρχοντα ενεργό Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια πολύ πιο υψηλή κινητικότητα, πολύ πιο έντονη στο μέλλον και θα είναι βεβαίως προς το συμφέρον της οικονομίας μας και των επαγγελματιών να υπάρχουν καταρτισμένοι εργαζόμενοι από τις χώρες μέλη μας. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες να αποτελούν ένα φραγμό, αντίθετα θα πρέπει να αποτελούν ένα σημείο κλειδί, μια απάντηση κλειδί στις προκλήσεις, τις οικονομικές και τις δημογραφικές. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα εκπαιδευτικά συστήματα στι χώρε μέλη μα και να το έχουμε υπόψη μα. Και επιτρέψτε μου, πριν ολοκληρώσω, να σα πω ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που γνωρίζω ότι πάρα πολλοί από εσά υποστηρίζουν, γιατί μου το έχετε αναφέρει και προσωπικά. Έχουμε να κάνουμε εδώ συγκεκριμένα με το θέμα τη επαγγελματική κάρτα της Πανευρωπαϊκής Επαγγελματικής ε, Κάρτα που θα αναφερθεί και στην ανακοίνωση μας, στην παρουσίασή μας αύριο για το ε, Single Market Act. Αυτή η κάρτα θα μπορούσε ανά επάγγελμα να προσφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία για την ε, αναθέρμανση της ενιαίας αγοράς. Αυτό βοηθάει και τους επαγγελματίες στην κινητικότητά τους σε διάφορες χώρες και στις μετακινήσεις τους σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, ώστε να ασκήσουν το επάγγελμά τους ελεύθερα σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίως αντικαθιστά τις γραφειοκρατικές απαιτήσει για διαφορά έγγραφα. Αντικαθιστά πολλά έγγραφα και ελαφρύνει κατά πολύ την γραφειοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τη, γιατί αυτή η κάρτα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στις αρμόδιε αρχές, επειδή θα τους επιτρέπει να έχουν άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε ουσιώδει πληροφορίε σε σχέση με το κάθε άτομο. Νομίζω ότι η κάρτα πρωτίστως διευκολύνει την επαφή, τη σχέση μεταξύ ενός επαγγελματία, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, με τις δυτικές αρχές, Τη περιφέρεια ή τη χώρα στην οποία πηγαίνει να σχέσει το επάγγελμα του, επιτρέποντα αυτέ τι χώρε να έχουν άμεση και γρήγορη πρόσφαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών που αφορούν τον επαγγελματίο αυτό. Η κάθε αυτή θα μπορούσε λοιπόν να συνδεθεί με μια βάση δεδομένων Ίσως το σύστημα IMI θα μπορούσε να αποτελέσει από αυτού ένα σημείο κίνησης. Πάντως θα είναι οπωσδήποτε χρήσιμο στις υπηρεσίες καταναλωτών ή εργοδοτών που μέσω της κάρτας θα ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ένα άτομο το οποίο είναι πλήρως καταρτισμένο. Αυτά, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι μια κάρτα επαγγελματική ε, που θα έχει τέτοιο χαρακτήρα θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τους επαγγελματίε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ε, συνεργάτες μας εδώ για την ε, υιοθέτηση της κάρτας αυτής και βεβαίως θα κάνουμε και επαφές και διαλόγους με τις επαγγελματικές οργανώσεις ξεκινώντας με τις οργανώσεις οι οποίες ήδη εξέφρασαν τη διάθεσή τους να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν μαζί μας για το θέμα αυτό. Αυτά είχα να πω Πρόεδρε. όσον αφορά τις σκέψεις μας και καταλήγοντας θα ήθελα να επαναλάβω κάποια πράγματα για να είναι σαφή. Πρώτον, το πρώτο αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταδεικνύει ήδη την ανάγκη εξυγχρονισμού της οδηγίας. Δεύτερον, σήμερα θα ακούσω προσεκτικά όλους αυτούς οι οποίοι ασχολήθηκαν με, την, με τον εξυγχρονισμό της οδηγίας. Τρίτον, η οδηγία και ο εξυγχρονισμός της προϋποθέτει κάποια διακυβευόμενα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Τέταρτον, η κάρτα και διαβούλευση με τις επαγγελματικέ οργανώσεις. Νομίζω ότι έχει έρθει πια η ώρα να περάσουμε από τις ιδέες στις συγκεκριμένε λύσεις. Πέμπτον, προβλέπω την έκδοση πράσινης βίβλου του χρόνου και το 2012 θα ακολουθήσει νομοθετική πράξη μετά από μελέτες, αντικτύπου κλπ. Αυτά σε σχέση με τις ε, θέσεις και τις πράξεις μας και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ σήμερα από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να με ακούσετε όσον αφορά την οδηγία. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Επίτροπε, σύντομα να πω, επειδή δεν έχετε χρόνο, ότι εξ ονόμας Επιτροπής και εξ ονόματος όλων αυτών που μετακινήθηκαν και ήρθαν να συζητήσουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την διαθεσιμότητά σας, για την παρουσία σας, για την ομιλία σας σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας. Ξέρετε πόσο και ευρωβουλευτές αλλά και εθνικοί βουλευτές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην, για την οδηγία αυτή και την αναθεώρησή της που νομίζουμε ότι είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάπτυξη, για την κατάσταση της ενιαίας αγοράς, για τους πολίτες και αλλά και για την ασφάλεια των ίδιων των επαγγελματιών. Έχω πει επανειλημμένως ότι είναι πολύ σημαντικό, μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης να ξαναβρούμε ένα δυναμισμό και είναι απαραίτητο να δώσουμε ελπίδα στους νέους επειδή η επαγγελματική επιτυχία διέρχεται και από την παραμονή στο εξωτερικό και από κατάρτιση που γίνεται στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν είχαμε μια πολύ καρποφόρα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και πριν να φύγετε θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια βασικά στοιχεία εδώ. Δηλαδή η κινητικότητα είναι απόλυτα ουσιώδης, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τις προϋποθέσεις της κινητικότητας αυτής και για τους νέους που καταρτίζονται και που χρειάζονται την κατάρτιση αλλά και για την νομική ασφάλεια που χρειάζεται και που αναγνωρίζουν και οι ίδιες οι επαγγελματικές οργανώσεις. Αναφέρθηκε ο κίνδυνος με στατιστικές οι οποίες είναι αόριστες, θα πρέπει να γίνει κάτι. βεβαίω η γλωσσική κατάρτιση αναφέρθηκε παρελειμμένως από πολλούς βουλευτές και επίσης εμείς εδώ θέσαμε το θέμα των της προσωρινής άσκησης επαγγέλματος κάτι το οποίο σημαντικό όσον αφορά την νέα-νέα αγορά και εδώ θα πρέπει βέβαια να βαθύνουμε τη σκέψη μας σε συνεργασία με τους εθνικούς βουλευτές. Μας δόθηκαν κάποιες ενδείξεις πολύ σημαντικές όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών διπλωμάτων. Μιλήσατε προηγουμένως για συνέπεια και διαφάνεια. Γιατί να μην συγκροτήσουμε λοιπόν μια ανεξάρτητη ε, ε, επιτροπή με συμμετοχή με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ανεξάρτητη λοιπόν επιτροπή με εμπειρογνώμονε, η οποία ε, δεν θα είναι αντικείμενο καμιά υποψίας ή καχυποψίας ώστε να υπάρχει ακριβώς ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Θα ήταν καλό να γίνει αυτό. Επίσης θέσαμε το θέμα της εναρμόνισης της κατάρτισης. Μιλήσαμε για την διαδικασία τη Μπολόνια, μιλήσαμε για τα όρια τη και μιλήσαμε για ένα θέμα της ε, εκπαίδευσης online. Δηλαδή η εναρμόνιση και η αναγνώριση που θα μας απασχολήσει σε αυτή την περίπτωση και βεβαίως αυτή η επαγγελματική κάρτα που γνωρίζω ότι είναι κάτι που για κάποια επαγγέλματα προχωράει πολύ γρήγορα και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να ισχύσει για όλους. Ποια θα είναι λοιπόν τα κριτήρια και πώς θα διασφαλίσουμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων είτε πρόκειται για τους πολίτες, τους καταναλωτές ή τους επαγγελματίες ακολουθώντας μια στάση έτσι ενεργητική και λαμβάνοντας υπόψη και κρούσματα όπως αυτό που αναφέρατε του Ισπανού γιατρού που δεν μπορούσε να ασχίσει το επάγγελμά του στην Ισπανία και πήγε στην Βρετανία. Αυτά Νομίζω ότι η συζήτηση που έγινε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο βέβαια, γιατί βρισκόμαστε ακριβώ στην καρδιά τη διαδικασία τη Λισαβόνα. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλους εσά. Και κύριε Επίτροπε, πριν αποχωρήσετε θα σα δώσω το λόγο για να κάνετε κάποια συμπεράσματα γνωρίζοντα βέβαια ότι εμεί μπορούμε να βασιστούμε σε εσά και εσεί σε εμά. Κυρία Πρόεδρε, μίλησα και πολύ αρχικά ε, και εσείς βεβαίως ε, ξέρω ότι χρειάστηκε να προσέξετε πολλούς σοβαρούς ομιλητές, γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Ε, συμφωνώ με την κινητικότητα αλλά πρέπει να λαμβάνουμε κάποια μέτρα, κάποιες προφυλάξεις ε, η κινητικότητα λοιπόν ναι αλλά υπό όρους και προϋποθέσεις και βεβαίω ε, αυτό δεν αφορά μονάχα τις επιχειρήσεις. Ε, όπως και η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά μονάχα τις επιχειρήσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε για συλλογική και για ατομική ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από κάθε περιφέρεια, πέρα από κάθε κοινότητα, πέρα από κάθε ε, χώρα ε, ε, που πρέπει να είναι ανταγωνιστικέ. Υπάρχει και ο, ο πολίτης της που πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Έχουμε τα εργαλεία των επαγγελματικών προσόντων, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον εργαλείο και η οδηγία αυτή μπορεί ε, να βοηθήσει τον έλεγχο ε, των, της κινητικότητας. Και βεβαίως η ενιαία αγορά, αυτή η μεγάλη ενιαία αγορά πρέπει να αποφέρει κάτι. Ε, και εγώ είμαι πολιτικός άνδρας και βρίσκομαι μεταξύ πολιτικών ανδρών και γυναικών, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα ερωτήματα ε, των μικρών επιχειρηματιών, των μεμονωμένων πολιτών που ρωτάνε και εγώ, εμένα τι θα μου προσφέρει, τι θα μου αποφέρει εν πάση περιπτώσει αυτή η Ευρώπη, αυτή η μεγάλη εσωτερική αγορά. Και εμείς θέλουμε να μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Προστασία, άνοιγμα προς άλλες αγορές, μια μεγάλη αγορά. Ε, δυνατότητα ε, καλύτερης κατανάλωσης, ε, ε, πιο εύκολη πρόσβαση στην κινητικότητα πολλά πράγματα. Θέλουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες να παρουσιάσουμε μια μεγάλη ενιαία αγορά που θα είναι η βάση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όσο καλύτερα λειτουργεί αυτή η βάση, αυτό το θεμέλιο, είτε πρόκειται για τοπικές, για περιφερειακές, για εθνικές, για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, μικρές, μεγάλες, ε, στρατηγική του 2020, ό,τι και να βάλουμε πάνω στο θεμέλιο αυτό θα βασιστεί σε σωστές βάσεις και επομένως θα αναπτυχθεί σωστά συνάδελφος Έγκον Κουίν που κάνει πολύ καλή δουλειά ε, για την έρευνα έχει αναπτύξει αυτήν ε, την ε, στρατηγική για το 2020 που, στην οποία θέτει ως προτεραιότητα την καινοτομία, την έρευνα και βεβαίως εκεί χρησιμοποιείται και το εργαλείο του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας εμείς θέλουμε να ε, ε, απεμπλέξουμε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γιατί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοστίζει 20 φορές παραπάνω για τις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από ό,τι σε άλλες ε, επιχειρήσεις σε άλλα σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν λειτουργήσει καλύτερη η εσωτερική αγορά λόγω ενός εύκολα επιτυγχανόμενου ευρωπαϊκού και καλά λειτουργούντος ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα λειτουργήσει καλύτερα όλη η αγορά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι που ήρθατε εδώ, που με ακούσατε με προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ ε, εκ των προτέρων για την, ε, για την συμμετοχή σας στον μεγάλο ε, ανοιχτό ευρωπαϊκό διάλογο που θα ξεκινήσουμε από αύριο για την Single Market Act και βεβαίως ε, πρέπει να πούμε ότι αυτή η ενιαία αγορά θα λειτουργήσει καλύτερα ε, και θα προστατεύσει καλύτερα τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις μικρές, τις μεσαίες ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομι... Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε ε, Επίτροπε Μπαρνιέ. Βεβαίω λειτουργεί καλύτερα η Ευρώπη και χάρη στον διαρκή διάλογο που έχουμε μεταξύ μας και στο διάλογο που έχουμε ε, με τους άλλους πολιτικούς φορείς ε, της Ευρώπης. Νομίζω ότι πραγματικά εάν λειτουργήσει καλά αυτή η ενιαία αγορά τότε μια πολύ μεγάλη πρόκληση θα έχει αντιμετωπιστεί ε, πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για αυτό το μεγάλο όραμα της ε, ευρωπαϊκής ταυτότητας και πιστεύω ότι τελικά, τελικά δεν θα, έχετε κανένα λόγο να άρχιστε να μας μιλάτε. Μα αστειεύομαι βέβαια, πάντα θα θέλουμε να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ ειδικά αυτούς που ήρθαν από μακριά για να μιλήσουν μαζί μας. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και είναι και αυτονόητο τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι εδώ και πολλούς μήνες εργάζονται έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αυτόν τον τραχή δρόμο της Ευρωπαϊκής ε, ηθαγένειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πρόκειται για ένα δρόμο που είναι μακρύς αλλά πιστεύω ότι πρώτον δεν θα είσαστε μόνοι σας, θα τον διανύσουμε μαζί, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως τα Εθνικά Κοινοβούλια και όταν θα πάτε στα εθνικά σας κοινοβούλια θα τους μεταφέρετε το μήνυμα ότι δουλεύουμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.